Okay, so, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε την απόψινη συνεδρίαση με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Αν δεν υπάρχει ένσταση, θεωρούμε λοιπόν ότι η ημερησία διάταξη έχει εγκριθεί. Ανακοινώσει του Προέδρου δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, εκτός του ότι έχουμε διερμηνία σήμερα σε 19 γλώσσες και όπως συνήθως ε, θα βρείτε και ηλεκτρονικά το αρχείο της συνάντησης. Και κάτι άλλο πιο σημαντικό, στις 9 Ιανουαρίου ακυρώνεται η συνεδρίαση που είχαμε προγραμματίσει και θα αντικατασταθεί από μια συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, εδώ στο Στρασβούργο, όπου είναι πολύ πιθανό έως και πιθανότατο θα έλεγα να είναι εδώ ο Τιερή Μπρετών για μια πρώτη ενταλλαγή απόψεων επί πολλών θεμάτων ε, αρμοδιότητας της ΕΝΒΗ και του χαρτοφυλακίου του Μπρετών. Πάμε στο άλλο σημείο τη ημερήσια διάταξη, ανακοίνωση του Πρόεδρου όσον αφορά τις συστάσεις των συντονιστών τη Δευτέρα Δεκεμβρίου που σας εστάλησαν ηλεκτρονικά όπως συνήθως, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Έχουν εγκριθεί. Πάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξης της απόψινης συνεδρίασης όπου στις 8 ε, και 10, 8 και 4 θα έχουμε την πρώτη ευκαιρία για μια πρώτη ανταλλαγή απόψε με τον Φραν Τίμερμαν για την Πράσινη Συμφωνία. Αλλά πριν από τι λύσει, έχουμε να ακούσουμε τα προβλήματα μαζί με εσά. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, ε, φιλοξενούμε εδώ τον Hans Μπρένεξ, ε, επικεφαλής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων, αλλά φυσικά θα εστιαστούμε λιγότερο στον ίδιο τον οργανισμό και περισσότερο στην έκθεση που εκδώσατε πριν δύο εβδομάδες περίπου και η οποία φυσικά είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ξεκινάμε με αυτό λοιπόν. Έχετε νομίζω και διαφάνειες, έχετε 10 με 15 λεπτά και μετά θα έχουμε την Γιούτα ε, για δύο λεπτά ως άτομο επαφή και μετά κάτσε για όποιον θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ σηκώστε χέρια σας για να σας καταγράψει η γραμματεία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ απόψε για να σας παρουσιάσω το περιεχόμενο της εκθεσής μας για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Δεν χρησιμοποιείται χαρτί, όπως ξέρω εδώ στην Επιτροπή, σας φέραμε ένα μικρό μικρό χαρτάκι, το οποίο θα βρείτε πάνω στα έδρανά σας ε, και περιλαμβάνει τον κωδικό QR και μπορείτε να κατεβάσετε έτσι την έκθεση στι συσκευές σας. Κάθε πέντε χρόνια ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος συγκεντρώνει τις καλύτερες γνώσεις ε, στην Ευρώπη για το κλίμα και τα σχετικά ζητήματα και πραγματοποιεί μια αξιολόγηση τη κατάσταση του περιβάλλοντο και τα συσχετίζει αυτά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για να παρακολουθεί κατά πόσο ε, είμαστε σε καλό δρόμο για του στόχου που έχουμε θέσει. Επίσης κοιτάμε μπροστά και μία δεκαετία, δεκαπενταετία για να διακρίνουμε τις τάσεις. Φυσικά αυτό δεν το κάνουμε από το πουθενά, αλλά σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και πρέπει να πω ότι την τελευταία πενταετία, μετά την τελευταία μας ε, έκθεση, το παγκόσμιο πλαίσιο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ε, προκλήσεις ε, άνευ αλλά και τεράστιες γνώσεις. Τα βασικότερα πάνελ, επιστημονικά πάνελ που εξετάζουν τα κλιματικά θέματα Μα στέλνουν τέτοια μηνύματα. Ξέρετε την έκθεση IPCC, το, την έκθεση του 1,5 βαθμού, του, την έκθεση για τους ωκεανούς. Ε, αυτές οι εκθέσει μας ενημερώνουν για τις αλλαγές στο κλίμα. Επίσης, ε, η έκθεση IPBES ε, είναι σημαντική, αφορά τι υπηρεσίε βιπικιλότητα και οικοσυστημάτων που αναφέρεται στην, σε τεράστια εξαφάνιση ειδών και επίση έχουμε και το Resource Panel που ασχολείται με τη χρήση των πόρων στον πλανήτη, πόσο βιώσιμη είναι η χρήση και πόσο μη βιώσιμη και πώ επιδρά το μοντέλο που χρησιμοποιούμε εμεί για τη χρήση πόρων στο κλίμα και στη βιοπικιλότητα. Όλα αυτά τα πάνελ καταλήγουν στα ακόλουθα τέσσερα συμπεράσματα. Πρώτον, για να αναστρέψουμε τι τάσει ε, χρειάζεται επιγόντω δράση. Και τα τρία πάνελ λένε το ίδιο. Δεύτερον, ήδη ζούμε σε εποχέ ε, μη αναστρέψιμες οι ζημιέ που έχουν γίνει δηλαδή δεν είναι αναστρέψιμε ε, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Τρίτον, αρχίζουμε να παρατηρούμε σημεία καμπής. Μηχανισμοί που επιταχύνουν, κλιμακώνουν αρνητικές τάσει και αποτελέσματα και πέραν αυτών επιπλέον αυτά τα τρία στοιχεία είναι αλληλένδετα. Επίσης, ε, είναι αλληλένδετα και σε διαστάση πολιτική, ε, όπω λέμε. Εάν αποτύχουμε σε ένα από τα τρία ε, σε μία από τι τρει πολιτικέ θα αποτύχουν και οι άλλε δύο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε θέματα ε, αλληλένδετων πολιτικών. Ποια είναι η κατάσταση τώρα του περιβάλλοντο στην Ευρώπη. Μιλάμε για την τάση τη τελευταία πενταετία δεκαετία. Ε, το ονομάζουμε το σχέδιο για το, ε, συγγνώμη, το πιάνο, της, ε, το, πλη, το, πιάνο για ευρωπαϊκού Περιβάλλοντο. Κάθε πλήκτρο του, πληκτρο, του πιάνου αυτού είναι μια πολιτική με δείκτε που αφορά μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Και αυτό που βλέπουμε σαφέστατα είναι ότι στη μέση του πίνακα αυτού παρατηρείται πρόοδος, μειώνονται οι εκπομπές άνθρακα και χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά οι πόροι. Αλλά άμα πάτε να δείτε το φυσικό κεφάλαιο, το συνολικό σύστημα, οι πιέσει ε, που ασκούνται πάνω στη φύση και στην βιοποικιλότητα είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε τις αρνητικές τάσει. Ε, βλέπουμε πιο αναμεικτή εικόνα για την ε, ανθρώπινη υγεία και τη φύση. Θα σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε αργότερα. Αν πάμε να δούμε πιο μπροστά προ το 2030 είναι σαφέ ότι το πράσινο εξαφανίζεται σιγά σιγά ως χρώμα και αυτό μας ε, λέει ένα σημαντικό μήνυμα ότι πρώτον δεν οφείλεται στο ότι δεν φέρνουν αποτελέσματα ευρωπαϊκές πολιτικές, οφείλεται στο ότι οι συνολικές συστημικές πιέσεις από την απώλεια πυκλότητα, από την κλιματική αλλαγή και από κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα επισημάνω δεν αντιστρέφουν τις τάσεις, διατηρούν τις αρνητικές πιέσεις στον πλανήτη μας και στις κοινωνίες μας. Αν πάμε δούμε το φυσικό κεφάλαιο, όπου τα πράγματα είναι τα χειρότερα, βλέπετε δύο πράσινες γραμμές. Εκεί έχουμε τις ε, καλύτερα προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 και άλλα συστήματα προστασίας και οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Αλλά άμα πάτε να δείτε τα άλλα στοιχεία, παρατηρούμε πρώτα απ' όλα στις τάσεις πρώτη ε, κυρίως ε, κόκκινο και ε, κίτρινο, αλλά άμα δούμε τους στόχους πολιτικής παρατηρούμε πολύ σημαντικό κενό υλοποίηση. Με τα βίας επιτυγχάνουμε τους στόχους ε, που έχουμε καθορίσει για το 2030. Η βελτιωμένη λοιπόν υλοποίηση και η συνεχής εστίαση στην υλοποίηση στα κράτη-μέλη και στους κλάδους από τους οποίους εξαρτώνται αυτά τα αποτελέσματα είναι κρίσιμη. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα ε, επικονιαστών. Ξέρουμε ότι αυτή είναι σημαντική για το διατροφικό σύστημα και οι πεταλούδες των λιμόνων ε, είναι πολύ σημαντική για τους ως επικονιαστές στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ε, μείωση 39% τα τελευταία 25 χρόνια. Αν πάτε να δείτε μετά πού έχουμε μετρήσει, καταμετρήσει αυτές τις πεταλούδες, ε, κυρίως σε γεωργικές περιοχές παρατηρούνται και το ίδιο βλέπουμε και για τα πουλιά ε, γεωργικών καλλιεργούμενων ζωνών, ε, τα αμφίβια και άλλα είδη που ευδοκιμούν εκεί. Αυτό μας δίνει μια ένδειξη της πίεσης στα οικοσυστήματα. Επιπλέον έχουμε τον κατακαιρματισμό του τοπίου, διαρκή συσσόρευση κάποιων ρήπων και κλιματική αλλαγή η οποία οδηγεί σε αρνητικές τάσεις στη βιοποικιλότητα. Αν σκεφτεί στην την κυκλική οικονομία ως βασικό στοιχείο για το μέλλον, εδώ και 12-13 χρόνια βλέπουμε πολύ χαμηλή αύξηση της κυκλικότητας. Ε, έχουμε εξετάσει, έχουμε πάει σε αυτή την περίοδο από 8 σε 12%, αλλά νομίζω ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι η πρώτη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα για να παρουσιάσει την ε, έννοια αυτή, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, να γίνουν κάποιε μετρήσει και να δοθούν και κάποια κίνητρα στου φορεί για να το υλοποιήσουν. Αλλά η πραγματική τάση ε, προ την κυκλικότητα δεν έχει ακόμα λάβει χώρα. Με αυτή την ταχύτητα δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουμε του στόχου του 2030 ή του 2050. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφάνεια. Μας δείχνει το επίπεδο φιλοδοξίας για το κλίμα. Τώρα βρισκόμαστε στο μείον 23% στην Ευρώπη, ενώ η οικονομία μας έχει σημειώσει αύξηση πάνω από 50%. Είμαστε δηλαδή η μόνη ήπειρο που έχει αποσυνδέσει πλήρως ε, ε, ε, επιτυχώς την οικονομία μας από τις εκπομπές ρήπων. Αλλά για να γίνουμε κλιματικά ουδέτερη ήπειρος, τα σχέδια και οι πολιτικές μας θα μας πάνε στο μείον 36% ή σε μείον 45% αν υλοποιούσαμε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, καλά σε εθνικό επίπεδο. Κανένα από αυτά τα δύο, ωστόσο, δεν θα μας οδηγήσει να γίνουμε η πρώτη ε, κλιματικά ουδέτερη η δηλαδή η συζήτηση του μείον 50, 55% είναι πολύ σημαντική, όπως καταλαβαίνετε, ε, παρατηρώντας αυτές τις τάσεις εδώ. Όσον αφορά τη σύνδεση όχι μόνο με την υγεία αλλά και με τη γενικότερη ρήμανση και την πίεση που ασκείται στα συστήματα, θα ήθελα να αναφέρω την πολιτική για τα χημικά. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, έχει τα καλύτερα συστήματα αξιολόγηση επικινδυνότητα χημικών στον κόσμο. Βασίζεται στον κανονισμό REACH κυρίω από την ΕΚΑ στο Ελσίνκι αλλά και από την ΕΦΣΑ, την αρχή ε, ασφάλεια των τροφίμων στην Πάρμα. Ε, είμαστε πρωτοπόροι. Αλλά αν δείτε τι πολλέ χιλιάδε χημικά που χρησιμοποιούμε στις οικονομίες μας, ελάχιστο ποσοστό το γνωρίζουμε τι πραγματικού κινδύνου ενέχει. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν εδώ είναι ότι για τη νέα πολιτική για τα χημικά ε, που δεν ε, κάναμε ε, πρόσφατα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο τομέας των χημικών είναι πολύ σημαντικός για να επιτύχουμε τους στόχους μας και να θεωρήσουμε ότι αυτός ο κλάδος θα πρέπει να κινηθεί προς την βιωσιμότητα, προς έννοιε όπως πράσινη χημεία ή ασφαλής, ασφαλού σχεδιασμού, κάτι που συζητείται αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που χρησιμοποιούμε εδώ το παγόβουνο. Κάποιες χώρες έχουν βάλει τα πιο επικίνδυνα χημικά του στο πέρμαφροστ, στι τρώσει του πάγου και καθώ αυτά λιώνουν, βλέπουμε να εκλείονται πολύ επικίνδυνα χημικά στα υδάτινα σώματα, στον ωκεανό. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτό το σχέδιο με το παγόβουνο εδώ. Μία από τις αποκρίσεις που έχουμε παρατηρήσει στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τα περίπλοκα ζητήματα διατομεακά, σε διάφορους τομείς όπου ασκούνται διάφορες πρακτικές που πλήττουν το περιβάλλον, είναι η ολοκλήρωση των πολιτικών. Ε, αυτή έχει μια ιστορία πάνω από 20 χρόνια, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα περίμενε κανείς. Αν δείτε τη χρήση αζότου στις αρρώσιμες, στις καλλιεργούμενες περιοχές που καταλήγουν στα ε, ύδατα της Ευρώπης, ε, και τώρα έχουμε περάσει από διάφορου κύκλους πρασινίσματο τη ΚΑΠ, αλλά οι συστημικέ πιέσει ε, στα γεωργικά συστήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώ από αυτό το πρασίνισμα και έτσι ασκείται πίεση στα υδάτινα σώματα, στην ποιότητα των υδάτων και στην βιοπικιλότητα, την υδάτινη βιοποικιλότητα κυρίω. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν, για να απαλύνουμε αυτέ τι πιέσει, θα χρειαστεί να κινηθούμε προ μια συστημική κατανόηση του πού πρέπει να ασκηθούν πολιτικέ και εργαζόμαστε με ένα μοντέλο όπου οργανώνουμε τι γνώσει μα σε τέσσερα συστήματα κλειδί. Το σύστημα ε, διατροφή. δεν θα πω το γεωργικό γιατί αυτό περιπλέκει πολύ τη συζήτηση και δεν την κάνει ιδιαίτερα επικοδομητική αν περιορίσουμε το τρόφιμα μόνο στην γεωργική φάση, το σύστημα των τροφίμων, ενέργειας, κινητικότητας και ε, αστικού περιβάλλοντος. Φυσικά αυτά είναι τα κρίσιμα ε, συστήματα της κοινωνίας που οδηγούν σε ευημερία, που μας έχουν βελτιώσει τα επίπεδα ε, διαβίωσης, αλλά θα πρέπει να οργανωθούν αυτά εντός των οικοσυστημάτων που έχουμε, δηλαδή πρέπει να μπούμε στην ουσία των κινητήριων δυνάμεων της βιωσιμότητας ή μη βιωσιμότητας. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα χρειαστεί να εξετάσουμε κάποια κενά πολιτικής, όπως η πολιτική για τα τρόφιμα, η γη και το έδαφος. Είχαμε πολιτικές στην Ευρώπη που έχουν αποτύχει και θεωρούμε ότι η γη είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς πραγματική ε, βιωσιμότητα και το τομέα των χημικών, όπου οι αρχέ ασφαλού σχεδιασμού για παράδειγμα, η μηδενική ρήπανση, θα αλλάξουν σίγουρα την ατζέντα. Είναι σαφέ επίση ότι εδώ δεν μιλάμε για μια ατζέντα που θα χαραχθεί από τον Περλεμό τη Βρυξέλλη, τα Άμστερνταμ, οποιαδήποτε πρωτεύουσα. Θα είναι μια ατζέντα που θα απαιτήσει κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων τη κοινωνία, των πόλεων και των κοινοτήτων μα. Η πράσινη εδώ καμπύλη είναι η αισιόδοξη πειραματισμό με νέε τεχνολογίε που βασίζονται σε έρευνε ε, και καινοτομίε ευρωπαϊκέ ε, και σχετικέ πολιτικέ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα για παράδειγμα, για να καταλήξουμε σε πιο σταθερέ και καλύτερε συνθήκε. Επίση, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ε, που υπάρχουν τα προσκόμματα, δηλαδή να σταματήσουμε να βελτιστοποιούμε τρέχοντα μοντέλα τα οποία θα οδηγηθούν σε αποσταθεροποίηση και σε σταδιακή κατάρριξη ορισμένων συστημάτων. Τεχνολογίε όπω ο, ε, ο ε, κινητήρα εσωτερική καύση, όπω και επιχορηγήσει που βλάπτουν το περιβάλλον. Ξέρουμε ότι αυτέ ήταν κάποιε από τι κάποια σημεία διαφωνία. Αν τα χαρτογραφήσουμε καλύτερα όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε στην έκθεσή μα, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πιο σωστά τι προποθέσει που θα αποτρέψουν κοινωνική και περιβαλλοντική ζημία η επιτάχυνση και η κλιμάκωση όχι μόνο λύσεων αλλά και τη ε, κατάργηση των μη βιώσιμων στοιχείων θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να επιτύχουμε του στόχου του 2030. Στη διαφάνεια εδώ βλέπετε το μεγαλύτερο κίνδυνο όπω τον έχουμε εντοπίσει εμεί. Για να επιτύχουμε του στόχου του 2030 σε πολλού κλάδου, αυτό θα πρέπει να γίνει με επένδυση σε σημερινά συστήματα και τεχνολογίε, αλλά βρισκόμαστε ε, σε οριακά κέρδη ε, αποδοτικότητα και ε, οποιοδήποτε οικονομολόγο θα σα πει ότι αυτά είναι, κοστίζουν πολλά και είναι επικίνδυνα. Θα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ε, θα οδηγήσουν μάλλον σε κινητοποίηση μέσων και υλικών και προσωπικού. Το να πάμε λοιπόν από υψηλό κόστος και οριακή αποτελεσματικότητα για να καταλήξουμε από αυτό σε ένα πραγματικά αποδοτικό σενάριο είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και το πιο δύσκολο για τα επόμενα χρόνια. Εδώ, σε αυτό το χαρτί, βλέπετε μια γενική εικόνα του ΟΕΠ ε, κατά κεφαλήν και βλέπετε και τα μέρη όπου έχουμε την χειρότερη ποιότητα αέρα και βλέπετε ότι σε μεγάλο βαθμό επικαλύπτονται αυτά τα δύο στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε ε, και για τη δίκαιη μετάβαση καλύτερα το πού εμφανίζονται αυτά τα ζητήματα. Εδώ βλέπετε απλά έναν χάρτη ε, από αυτούς που έχει η έκθεση γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι στην Ευρώπη 25 και παραπάνω χρόνια από τότε που έπεσε το σύνδρομο παραπέτασμα ε, έχουμε ένα νέο σύνδρομο παραπέτασμα που χωρίζει την Ευρώπη σε πιο μολυσμένη και λιγότερη. Αυτό παρουσιάζουμε στην έκθεση και τελευταία διαφάνεια πιστεύω ότι η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτον, θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στην υλοποίηση. Το κενό υλοποίηση, το χάσμα υλοποίηση σε πολλέ πολιτικέ είναι τεράστιο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα λοιπόν καλύτερα. Το δεύτερο είναι ότι ε, αν συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στι υπάρχουσες προσεγγίσει πολιτική αποκλείται να φτάσουμε και να επιτύχουμε τις φιλοδοξίες ε, της Πράσινης Συμφωνίας ε, του 2030. Χρειαζόμαστε πιο συστημική βιωσιμότητα στις πολιτικέ μα. το τρίτο στοιχείο υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να γίνουν λάθο επενδύσει και να μα οδηγήσουν σε αδιέξοδο αντί σε καινοτομίε. Και επίση χρειαζόμαστε νέε θέσει εργασία και ανταγωνιστικότητα για το μέλλον σε όλη την Ευρώπη. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν μόνο από το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και το δυναμικό των κοινωνιών μα στο σύνολό του. Αυτό περιλαμβάνει επιχειρήσει, πολίτε ε, τη πόλη μα και αγροτικέ περιοχέ όπου υπάρχει τεράστιο ε, δυναμικό καινοτομία. Και αν εστιαστούμε και τα οργανώσουμε όλα αυτά καλά, θα είμαστε η πρώτη ήπειρο ε, που θα κινηθεί προς την ε, θεμελιώδη σημασία ε, κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της κλιματικής ουδετερότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Γιούτα Πάουλους, που είναι ο σύνδεσμός μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπρόνινγκς που ήρθατε απόψε και μας παρουσιάσατε το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής με τόσο εύληπτο τρόπο. Δεν κατάφερα να διαβάσω όλη την έκθεση, αν και κοίταξα τα κυριότερα σημεία στις Βρυξέλλες. Η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και Όποιος δεν έχει τι να κάνει τα Χριστούγεννα νομίζω πως εδώ θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να μάθει πολλά. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα της γνώσης πολλών έγκριτων επιστημόνων και θέλω να τονίσω ότι πολλά από τα στοιχεία, ειδικά για την βιωσιμότητα, έχουν συλληφθεί από εθελοντές. και ίσως γνωρίζετε πως υπάρχουν κόκκινες λίστες στην Ευρώπη, δηλαδή απειλούμενα είδη στο χείλος της εξαφάνισης. Θα πρέπει λοιπόν να μην στεκόμαστε μόνο στα απειλούμενα είδη, αλλά να ε, κοιτάζουμε και τα κοινά ε, είδη χλωρίδας και πανίδας. Υπάρχει Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάλλον να δούμε ότι από τη στιγμή που εξαφανιστεί ένα είδο τελείωσε. Αυτό είναι, δεν ξαναγυρίζει πίσω. Νομίζω πως η εκτίμηση αντικτύπου που θα γίνει εν ώψη της καινούργιας νομοθεσίας θα πρέπει να έχει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, αυτή η... αυτός ο σχεδιασμός με γνώμονα την ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικός και στην βιομηχανία χημικών προϊόντων. Υπάρχουν ορισμένες χημικές ουσίες, για παράδειγμα, που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Κάποιες ουσίες που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν ως αναπληρωματικά στρογόνα, για παράδειγμα. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν σφαιρικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα ως ε, κατευθυντήρια γραμμή. Νομίζω πως ε, πρέπει να είναι γνωμονάς μας η βιωσιμότητα και πρέπει να εξετάσουμε όλες ε, τις ε, πτυχές της σχετικής νομοθεσίας με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Θα ήθελα λοιπόν στην επόμενη περιβαλλοντική έκθεση να δω αυτά τα κίτρινα σημεία να έχουν αλλάξει χρώμα και να ξαναγίνουν πράσινα στους πίνακες που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Γιούτα, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω πως το μήνυμα που στέλνετε είναι ισχυρότατο και επίκαιρο. Η Νέα Πράσινη Συμφωνία παρουσιάστηκε και παρουσιάστηκε για πολλούς τομείς και θα σίγουρα θα μας απασχολήσει τα ερχόμενα χρόνια. Ακούσαμε μεγάλη προσοχή την παρουσίασή σας, ιδιαίτερα όταν αναφερθήκατε στα διάφορα χημικά και στο πού τραβάμε αυτή τη γραμμή μεταξύ του γεωργικού τομέα και το πώς επηρεάζει διάφορα είδη εντόμων, για παράδειγμα, και από την άλλη τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα φυτοφάρμακα και τα ζυζανιοκτώνα. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε και θα ήθελα περισσότερες ε, λεπτομέρειες και σίγουρα θα είμαι από αυτούς που θα διαβάσουν την έκθεση τα Χριστούγεννα. Επίσης, ε, έχω μια ερώτηση σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Συμφωνώ με τη Γιούτα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και να πω εδώ ότι όταν ήρθα στον οργανισμό σας πριν από κάνα δύο χρόνια, Συζήτησα μεταξύ ε, σας τι ανησυχίε των πολιτών για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και το πώς αυτοί επηρεάζουν τη γονιμότητα. Νομίζω πως εδώ νομιζω πω εδω χρειαζεται να αυξήσουμε τα επίπεδα της προστασίας, διότι δεν είναι μόνο το οικοσύστημα σημαντικό, αλλά και η υγεία των πολιτών. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι υπάρχει διασύνδεση ενδοκρινικών διαταρακτών και κοινών νόσων, από τις οποίες πάσχουν οι πολίτες της Ένωσης. Και να είστε σίγουρος πως ε, θα διαβάσω οτιδήποτε σχετικό στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φρόνιξ για την παρουσίαση. Ε, θα ήθελα να επανέλθω λίγο σε αυτή τη διαφάνεια που δείξατε για τι πεταλούδε, αν μπορείτε. Έχω ένα πρόβλημα με τα νούμερα που αναγράφονται εκεί. Εγώ βρήκα μια επιστημονική μελέτη για τις πεταλούδες στη Φλάνδρα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι οι πεταλούδες είναι αντικείμενο μελέτης από το 18ο αιώνα ακριβώς γιατί είναι τόσο εντυπωσιακέ. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία. Αν λοιπόν δούμε τι γίνεται στη Φλάνδρα θα το χαρακτηρίσουμε ως καταστροφή. Και γιατί αυτό. Διότι χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα αποτελεσματικές μεθόδους ε, γεωργικές, ψεκάζουμε χιλιάδες χιλιόμετρα με φυτοφάρμακα και ασκούμε τεράστια λοιπόν πίεση στο περιβάλλον. Και ως αποτέλεσμα οι πεταλούδες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ε, αυτό βέβαια ίσως θα ήταν μια ερώτηση για τον Μπάς και όχι για σας, αλλά ας περάσουμε λίγο ε, στην... στη βόρεια Βραβάντη και ε, στη χειροτροφία. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν, υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, χείρων σε αυτήν την περιοχή και νομίζω πως αυτό έχει επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν μπάσε σου δίνω δουλειά για τους επόμενους μήνες. Okay, Mr. for EPP.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 Citizen science was mentioned, volunteers. In, we call it citizen science. Αναφερθήκατε λοιπόν στους ε, εθελοντές ε, και για την ε, συλλογή στοιχείων. Οι εθελοντές είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Έχουμε εθελοντές, ορνηθολόγους, εντομολόγους, οι οποίοι μας βοηθούν πάρα πολύ. Και μάλιστα τρέχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προγράμματα με τη συνεργασία ε, διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και σε αυτό οφείλουμε λοιπόν τα πολυάριθμα στοιχεία που έχουμε. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, χρησιμοποιούμε διάφορες εφαρμογέ ε, σε κινητά τηλέφωνα που μπορούν να βοηθήσουν έναν απλό ε, πολίτη να κάνει τις δικές του μετρήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την γεωργία και την επισητιστική βιομηχανία. Νομίζω πως μπορώ να το πλαισιώσω διαφορετικά. Όμως ε, μπορώ να σας εξηγήσω γιατί χρειάζεται συστημική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία τροφίμων. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τέσσερις φορές το φαγητό μας. Πληρώνουμε ως αφορολογούμενος για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, το οποίο φαίνεται περίεργο γιατί ε, είναι αδιανόητο εκείνοι που παράγουν το φαγητό μας να μην μπορούν να κερδίσουν αρκετά χρήματα. Έπειτα, φυσικά πληρώνουμε όταν αγοράζουμε το φαγητό και σπάνια αγοράζουμε γεωργικά προϊόντα. Αγοράζουμε έτοιμη τροφή που έχει μεταποιηθεί, έχει προσθεθεί αλάτι, ζάχαρη. Δεν αγοράζουμε την πρώτη ύλη, το οποίο σημαίνει ότι πληρώνουμε μια τρίτη φορά ως φορολογούμενος για ε, τις ε, κλιματικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της επιστημιστικής βιομηχανίας και μια τέταρτη φορά όταν καταλήγουμε στο γιατρό, διότι το σύστημα παραγωγής τροφίμων δεν είναι υγιές είναι ασφαλές αλλά δεν είναι υγιές. Είμαστε λοιπόν στον 21ο αιώνα και νομίζω πως <coughs> μπορούμε να τα πάμε καλύτερα σε ό,τι αφορά ε, το φαγητό και την παραγωγή αυτού. Γι' αυτό και στην έκθεση ασχολούμαστε και με αυτές τις πτυχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά με τα χημικά και τον αντίκτυπο που έχουν σε τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην υγεία. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι πάνω από 620.000 ε, ανθρώπων πεθαίνουν πρόωρα λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά είναι στοιχεία ε, που διασταυρώνονται και με τον ε, ΠΟΗ. Επίσης, τα χημικά και η μόλυνση και η πολιτική σχετικά. Συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων. Γι' αυτό και φαντάζομαι πως οποιαδήποτε πολιτική προκύψει θα αφορά όλους. Γι' αυτό θα πρέπει αυτοί οι τρεις οργανισμοί να συνεργαστούν, τουλάχιστον αυτοί οι τρεις, έτσι ώστε να εκπονούν μία διετή, ας πούμε, η τριετή έκθεση σχετικά με τα χημικά. Υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχουν τα νούμερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η εντολή για κάποια από αυτές τις υπηρεσίες να κάνει αυτή την ενέργεια. la mejor ξέρω εγώ σε διάφορες περιοχές των κρατών μελών ξέρω ότι υπάρχουν ε, διάφορες ε, ελλείψεις, διότι υπάρχει έλλειψη σχεδίων διαχείρισης εκ μέρους της Κομισιόν. Μετά λοιπόν από την ε, ε, ίδρυσή τους αυτών των project, των προγραμμάτων, ακόμη έχουν μείνει στα χαρτιά. Από ό,τι είδα λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, Υπάρχει ανησυχία. Όλα αυτά λοιπόν τα πράσινα, τα μέρη εδώ, μέχρι το 2020, πιστεύετε ότι επειδή αφορά ε, περιοχές Natura και επειδή δεν γίνεται τίποτα και δεν εφαρμόζεται η οδηγία για το Habitat, δεδομένου ότι έχουμε και κάποιες πολύ ευαίσθητες περιοχές, τι θα γίνει. Όσον αφορά επίσης τα δάση και την δασική πολιτική που είναι θεμελιώδους μασίας για την Ευρώπη, διότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αποψηλώνουμε ε, παλιά δάση και να κάνουμε βιομηχανικές ε, περιοχές οι οποίες κάνουν εντατική δουλειά, καμιά φορά εκμεταλλεύονται και το προϊόν των δασών, κάνουν χαρτί και έτσι τα χάνουμε για πάντα αυτά τα δάση. <coughs> Sorry, for renew, Mr. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ευχαριστώ ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα πολύ καλά σχόλια και τις ερωτήσεις, αλλά δείξατε μία διαφάνεια που δείχνει κάποιο νεφιάλτη που έρχεται από το πρώην Σοβιετικό μπλοκ, το νέο νέφος, το οποίο εξαπλώνεται πάνω από την Ευρώπη. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα. Κάτι που συζητούν τα κράτη-μέλη, αλλά φαίνεται να μην έχει αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η καύση ανθρακά τόσο στη θέρμανση οικειών αλλά και στα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια αλλά και στις μεταφορές. Τώρα, εγώ αυτό που διερωτώ με είναι πέραν της δίκαιης μετάβασης. Υπάρχει κάτι πιο δύσκολο που θα οφέρεται στο γεγονός αυτά που δεν ακούμε. Ότι τα ευρωπαϊκά επίπεδα αποδεκτής ε, ποιότητας αέρα βασίζονταν σε συστάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Και αυτό είναι ο χαμηλότερο παρονομαστή, όχι η υψηλότερη ποιότητα. Ο, εγώ θα ανέμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η καλύτερη. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι θα ήταν ε, το διάγραμμα αυτό αν εφαρμόζατε το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε, κύριε Σκόκαλη, για την ΚΟΕ. thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για την έκθεση. Θα το διαβάσω τα Χριστούγεννα. Προσθέτει πολλές πληροφορίες ε, στην παγκοσμία γνώση για την καταστάση του περιβάλλοντος, όπου δεν υπάρχουν σύνορα φυσικά. Αυτή η εκθέση προέρχεται από το δικό μας οργανισμό και υποχρεούμεθα όλοι να συμβάλλουμε στην επιστήμη και να παράγουμε πολιτική βάσει των κανόνων διαφωτισμού και την επιστημονική μεθόδου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη διαφάνεια με το πιάνο δεν πρέπει να το αφήσετε να παίξει αυτό το πιάνο ένα ρεκδιέμ, διότι δεν θα είναι ρεκδιέμ του περιβάλλοντος ή του πλανήτη, είτε για τους χείρους είτε για τις πεταλούδες, θα είναι για την ανθρωπότητα. Ε, climate security is the ultimate human. Και η κλιματική ασφάλεια είναι το απότερο ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορούμε να μηνύσουμε εδώ το πιανίστα, γιατί εμεί είμαστε οι πιανίστε. Είναι δική μα δουλειά να προστατεύσουμε τον πλανήτη και μπροστά μα. Έχουμε 30 δράσει κλειδιά, σημεία πολιτική που είναι αναγκαία, ώστε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να γίνει επιτυχία. για να κάνουμε όλα αυτά τα πλήκτρα πράσινα, αντί για κόκκινα. Και όπω γνωρίζετε από χθε, θα πρέπει να ασχοληθούμε προσωπικά, να εργαστούμε και να καθοδηγήσουμε τον κόσμο προ την κλιματική ασφάλεια και την κλιματική δικαιοσύνη. Οπότε η ερώτησή μου προ εσά κύριε Δευθυντά, αυτές τις εποχές ε, έκτακτης ανάγκης. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να διαθέσουμε αυτές τις παρουσίες, αυτά τα δεδομένα περισσότερο στους πολίτες, στους επιστήμονες, στους πολιτικούς ε, και πιο συχνά αντί για κάθε πενταετία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Christensen. Ευχαριστώ κύριε Κρίστιανσεν. Ευχαριστώ, θα μιλήσω δανέζικα. Yes. For mig kan og skal øh, intensiv landbrug gå hånd i hånd Από όσο ξέρω εγώ, η εντατική γεωργία πρέπει να κινείται παράλληλα με τη βιοπικιλότητα. Δέκα δισεκατομμύρια θα είναι η, σύντομα η κάτοικοι του πλανήτη. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο θα συνδυάζει την εντατική γεωργία και τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αυτό και στην ΚΑΠΑ και στην Πράσινη Συμφωνία. Να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να δράσουμε για βιώσιμη γεωργική παραγωγή. Ε, Η κυρία Ελεονόρα Εύη, παρακαλώ, είμαι εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ιταλικά. Δύο ερωτήσεις ήθελα να σας κάνω. Η πρώτη είναι ένα θέμα που αναφέρατε προηγουμένως στο έδαφος. Διότι και από την εκθεσή σας προκύπτει ότι οι συνθήκες του εδάφους δεν φαίνεται να είναι καλές, δυστυχώς. Με στην τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, έχουν επιδεινωθεί δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε. Και γνωρίζουμε δυστυχώ και του λόγου που οδήγησαν στο να μην εγκριθούν και δεν υπάρχουν σχετικοί ευρωπαϊκοί στόχοι. Και ήθελα να σα ρωτήσω αν στο πλαίσιο αυτή τη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσεί θα προτείνατε να προταθεί ένα στόχο ουδετερότητα όσον αφορά την υποβάθμιση του εδάφου μέχρι το 2030. Και μετά άλλη μια ερώτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την καύση, την αποτέφρωση των απορριμμάτων, διότι πρόσφατα είδαμε μια μελέτη σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία μαζί με τον συντονιστή του Ιταλικού Κέντρου για το Περιβάλλον, έδειξε αυτή η μελέτη ότι σήμερα η δυνατότητα αποτέφρωση των απορρίμματων στη δική μου χώρα, στην Ιταλία, αντιστοιχεί σε 13 ε, εκατομμύρια τόνους ετησίως. Με αυτό το ποσό μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα τα υπολοιματικά απορρίμματα που είναι 9,9 ε, τόνοι. Αυτά προέργαμε εμείς ε, πέρυσι. Οπότε αφού υπάρχει δέσμευση μείωση, πρόληψη και ανακύκλωση ε, για τα απορρίμματα, θέλω να πείτε εσεί ε, πώ κρίνετε την πίεση ορισμένων λόμπι που επιμένουν να κατασκευαστούν νέε εγκαταστάσει αποτέφρωση που σήμερα, κατά την άποψή μου, είναι μια ε, απερχαιωμένη πια πρακτική. Ευχαριστώ. And the last... Ε, και τέλος, η Grace O'Sullivan έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπρένιγκς για την παρουσίαση. Η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς που είμαστε υπεύθυνοι της πολιτικής. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ε, το εξή. Οι φυστάμενες προτάσεις για το πολιτέστημιο ουσιονομικό πλαίσιο εντάσσουν την, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη κατηγορία η οποία θα δεχτεί 14% μείωση προϋπολογισμού. Και η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς αυτό θα επηρεάσει τη δουλειά σας. Πώς θα μπορείτε μετά από αυτή τη μείωση να συνεχίσετε να παρέχετε αυτές ε, τις σημαντικές πληροφορίες και να ε, κάνετε όλα αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω το όνομά μου στον κατάλογο των ομιλητών. Αυτά είναι τα προνόμια του Πρόεδρου. Να επανέλθω λοιπόν στη διαφάνειά σας για τους διάφορους στόχους ε, μείωσης διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει κάποια οικονομική ανάλυση σχετική για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους. Διότι ο Φραντ Τσίμερμαν θα έρθει όπου να είναι, ε, αλλά αυτό είναι το ακόλουθο. Ποιος θα είναι λοιπόν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ε, με βάση αυτά τα νούμερα που βλέπουμε στις οθόνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω σύντομα. Λοιπόν, έγιναν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία για εύλογους λόγους. Νομίζω πως από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την ε, Πράσινη Συμφωνία δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη ευθυγράμμιση. Υπάρχουν οργανισμοί όπως ο δικός μας ε, οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία που έχουμε από την ε, επιστήμη. Ποτέ λοιπόν δεν υπήρχε τέτοια ευθυγράμμιση οργανισμών και επιστημονικών στοιχείων. Τώρα, αν εμεί έχουμε κάποια σχέση με τη διαδικασία, ναι, έχουμε, διότι συνεργαζόμαστε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν, με τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα και ήδη έχουμε έρθει σε επαφές με το επιτελείο του Φραντ Τίμερμαντς. Ε, συνεργαζόμαστε και με την ε, διεύθυνση ΜΑΡΕ και με την ε, διεύθυνση MOVE, με όλες αυτές τις σχετικές υπηρεσίες της Κομισιόν, έτσι ώστε να πλαισιωθεί το λεγόμενο MRV, ο έλεγχος δηλαδή και η επαλήθευση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά μόνο ε, κάτι για το οποίο έχεις στοιχεία. Και νομίζω πως ε, η Πράσινη Συμφωνία θα χρειαστεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν μετρήσεις και εδώ βρίσκεται ε, ο οργανισμός μας και η σημασία αυτού που κάνουμε. Τώρα, κύριε Γκοντζάλες, Νομίζω πως ε, μπορώ να σας απαντήσω λέγοντας ότι ήδη έχουμε εκπονήσει την ε, έκθεση που εξετάζει την καταλληλότητα των σχετικών οδηγιών για την προστασία της φύσης και αυτό έχει επιπτώσεις και ε, στις προστατευόμενες περιοχές και στις μη προστατευόμενες. Έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν μεν Υπάρχει μεν πρόοδο, όμως ε, υπάρχουν ελλείψεις στον σχεδιασμό. Χρειάζεται λοιπόν ο κατάλληλος σχεδιασμός με τους κατάλληλους πόρους και πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα προσωπικού, προβλήματα οικονομικής φύσεως. Επίσης, αρκετοί κάνατε ερωτήσεις για τη χρήση της γης στην ε, δασοπονία και τη γεωργία. Έχω να σας πω ότι δεν θα κερδίσουμε τη μάχη για τη πλότητα στο 20% της επικράτειας ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο το 20% της επιφάνειας του πλανήτη. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι πάνω από την ε, μισή επιφάνεια της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι στη θάλασσα. Και αν μετρήσουμε σε ναυτικά μίλια, είναι τεράστια η έκταση που πρέπει να προστατευθεί. Α μην ξεχνάμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση, διότι η βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα εκεί, όσο ρευστό είναι και το νερό. Μετά, ε, αναφερθήκατε στη δίκαιη μετάβαση, στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη, στο πρόβλημα του νέφους. Σας έδειξα στη διαφάνεια αυτή το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το διερευνήσετε περισσότερο, να δείτε τι, σημαίνει, τι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις και ποια είναι η διαφοροποίηση στα διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί με ε, την δίκαιη μετάβαση και θέλουμε να επενδύσουμε σημαντικά ποσά, θα χρειαστεί να κάνουμε ελέγχους, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ε, τα δεδομένα είναι καλά για πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο έλεγχο είναι επίση καλός, κανεί όμω δεν έχει ούτε την εντολή ούτε του ε, διαθέσιμου πόρους για να συνδυάσει αυτέ τι προσπάθειες. Η Eurostat και ορισμένοι άλλοι θα μπορούσαν ίσω να αναλάβουν αυτό το καθήκον, αλλά χρειάζονται εντολή. Θα ήθελα όμως να σας δώσω ένα παράδειγμα προς μίμηση που θα σας φανεί παράξενο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, εισήγαγαν περιβαλλοντική νομοθεσία πριν από περίπου 20 χρόνια. Γίνεται μια ετήσια έκθεση για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη η οποία βασίζεται σε στοιχεία. Μπορώ λοιπόν να φανταστώ τη δημιουργία ενός παρόμοιου μηχανισμού στην Ευρώπη, ο οποίος θα αναλύει τα προβλήματα, τις συνέπειες και τις νευραλγικές περιοχές. Και στην έκθεση αυτή θα, μπορούσε, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία για την ποιότητα του αέρα, όπως είπατε και εσείς. Τώρα, περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην Πρατισλάβα πριν από μερικές εβδομάδες ε, διεξήχθη το περιβαλλοντικό φόρουμ. Έχουμε ορισμένε ιστοσελίδε για την ποιότητα του αέρα όπου μπορεί να κάνει κλικ σε όποια πόλη τη Ευρώπη ε, θέλει και να διαβάσει τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα του αέρα. Μπορείς να δεις τα στοιχεία της ποιότητας του αέρα των περασμένων 100, των προηγούμενων 100 ημερών. Και νομίζω πως ε, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μείωση των θανάτων, αν χρησιμοποιήσουμε καλά αυτά τα στοιχεία. Πάνω από 140 ανθρώπους κάθε χρόνο μείωση. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Επίσης, ε, η ερώτηση με το πιάνο και τον πιανίστα. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Αυτό μας δείχνουν οι τάσεις. Αν όμως θέλουμε να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και αν υπάρχει και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων για το ποια θα είναι η πράσινη πρωτεύουσα, αν δηλαδή εφαρμόσουμε και υλοποιήσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας, φυσικά και μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον και μπορούμε, το μέλλον και μπορούμε να δούμε αυτά τα χρώματα να αλλάζουν, να γίνονται πράσινα. Ο πλανήτης μας λέει πως ε, πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε και να προσαρμοστεί η πολιτική μας στις νέες συνθήκες. Τώρα, τα δεδομένα μας θα ε, μπορούν να είναι διαθέσιμα στους πολίτες. Ναι, φυσικά. Υπάρχουν αρκετοί που παρακολουθούν τα στοιχεία αυτά, που μπορούν να χειριστούν και την τεχνολογία και πριν από ε, λίγα χρόνια είχαμε τρία εκατομμύρια μόνο ε, χρήστες. Τώρα αυτός ο αριθμός έχει υπερπολαπλασιαστεί. Φτάνουμε λοιπόν πιο κοντά στους πολίτες και χάρη στις επενδύσεις στο πρόγραμμα Κοπέρνικος που μας δίνουν γεωγραφικά δεδομένα που είναι εύκολα αντιληπτά από τους πολίτες γιατί είναι άμεσα ορατά, μπορούμε να βελτιώσουμε λοιπόν την ορατότητα και την απήχηση της δουλειά μας. Μετά, επισητιστικό σύστημα, παραγωγή τροφίμων, φυσικά και συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων αλλά όχι μόνο ο γεωργικός τομέας, αλλά και η αλία θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να, παράγει, να παράγονται τρόφιμα που είναι ασφαλή, που δεν ασκούν εξωτερικές ε, πιέσεις, ε, δεν επηρεάζουν τις τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει με τη Σόγια και που προφυλάσσουν το περιβάλλον, έτσι ώστε να μην το επιβαρύνουν. Και εδώ να απαντήσω και στην ερώτηση για τη γη. Αυτό που ζητάμε τώρα είναι η γεωργία που προστατεύει το περιβάλλον, η γεωργία που φροντίζει τη γη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ε, με καινοτόμες μεθόδους, είτε με εκτεταμένη γεωργία. Εμείς όμως πρέπει να δώσουμε το κίνητρο για να αλλάξει η κατάσταση. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε η στρατηγική από τη φάρμα στο πιάτο. Μετά, φυσικά και η γη υφίσταται πιέσεις και το χώμα και ο κατακαιρματισμός του φυσικού τοπίου και η αρπαγή της γης και όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν επιβαρύνει ε, το χώμα τα τελευταία 25 χρόνια. Σίγουρα είναι αντίθετες στους στόχους. Θέλουμε την επιστροφή της Αιγής στην αρχική της κατάσταση. Αλλά από όσο καταλαβαίνω, στους κύκλους πολιτικής γίνεται λόγος για αυτήν την αλλαγή. Επίσης, ε, να σας πω ότι θεωρώ πως η γενικότερη αρχή που πρέπει να διέπει την πολιτική είναι ε, το να υπάρχουν καλύτερα, ισχυρότερα οικοσυστήματα και η διαχείριση να είναι επίσης βελτιωμένη. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες είχα δει και ένα αυτοκόλλητο σε ένα αυτοκίνητο από πίσω μια φορά που έλεγε πρέπει να σταματήσουμε να φερόμαστε τόσο άσχημα στη γη. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Ε, και να περάσω στον προϋπολογισμό. Πράγματι, με την υφιστάμενη πρόταση υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται εντό εισαγωγικών σταθεροί σε ονομαστική αξία. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι θα γίνουν περικοπές η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα οδηγήσει σε 14% μείωση της χρηματοδότησης των οργανισμών αυτών. Υπάρχουν όμως ε, πάγια έξοδα, όπως ε, εκτηριακά, αμοιβέ ε, προσωπικού κτλ. για να καταφέρουμε να πιάσουμε αυτό το στόχο των περικοπών θα πρέπει να απολύσουμε το 20 του προσωπικού μας. Και αυτό είναι τελείως αντίθετο με τις προσπάθειες που γίνονται και με, για την Πράσινη Συμφωνία. Φυσικά και υπάρχει θέληση, θέλουμε να στηρίξουμε την ε, Πράσινη Συμφωνία με ό,τι κάνουμε, και, αλλά ελπίζω και ο προϋπολογισμός να συμβαδίσει με τους νέους στόχους πολιτικής. Είμαστε βέβαια ένας πάρα πολύ μικρός οργανισμός σε σχέση με άλλους. Έχουμε 210 υπαλλήλους, είμαστε, έχουμε πολύ μικρό budget και δεν ζητάμε εκατοντάδες νέες θέσεις για να αυξήσουμε τις ικανότητές μας, αλλά θέλουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την πολιτική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και ε, στην ε, Κομισιόν. Χρειάζεται όμως να στηριχτούμε για να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε με τη σειρά μας τα θεσμικά όργανα. Έπειτα, υπάρχουν στοιχεία για μία αξιολόγηση μακροοικονομική. Να δούμε τι θα γίνει με αυτές ε, τις ετάσεις που παρατηρούνται το μείον 45%, μείον 55%. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για ορισμένους κλάδους, για τις επενδύσεις για παράδειγμα, έχουμε αρκετά στοιχεία για τον τομέα της κινητικότητας, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η Πράσινη Συμφωνία. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αν συγκεντρώσουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν και συνδυαστικά τις χρησιμοποιήσουμε. Και φυσικά με τα χαράς θα συνεργαστούμε ε, με όσους θα εκπονήσουν την εκτίμηση αντικτύπου. Αλλά ας μην ξεχνάμε την κοινωνική, την ε, κοινωνικο-οικονομική διάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε διάφορα στοιχεία και δεδομένα έτσι ώστε να δούμε ολιστικά το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε εμένα τα συμπεράσματα τώρα όλη συζήτησης συζήτηση για δύο λεπτά από την κυρία Λένα, ναι, είμαι μέλος της ε, Διοικητικού Συμβουλίου και σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εργάζομαι καθημερινά ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λούντ. Η εργασία που παρουσιάστηκε σήμερα είναι πολύ σημαντική για να δημιουργήσουμε δυνατότητες στην Ευρώπη για να εφαρμοστεί η Πράσινη Συμφωνία. Το δυνατό σημείο του οργανισμού είναι τα ε, δεδομένα, η γνώση, η τεχνογνωσία, ό,τι έχουν όσον αφορά τα θέματα για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υποφάσει στην Ευρώπη. Επίσης, τα δίκτυα τα οποία έχετε στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά για όλα τα κράτη-μέλη. Ο οργανισμός είναι πολύ μικρός, όπως είπατε και προηγουμένως, αλλά σε σχέση με όλα τα θέματα που θα θέλαμε να καλύπτουμε. Και, και εκτιμούμε το γεγονός ότι συνέχεια ασχολείστε με νέα θέματα και αφήσαμε κάποια νέα θέματα την ε, ε, βιώσιμη χρηματοδότηση, τα είδη διατροφής λοιπά Ο ε, οργανισμός αναπτύσσει τη νέα τη στρατηγική για την επόμενη δεκαετία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει στο μέλλον. Θα ήθελα όμως να προσθέσω άλλη μία επιθυμία μου σε αυτόν τον κατάλογο, διότι μας παρουσιάσατε σήμερα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να δω εκθέσεις ετήσιες και αναφορές ετησίως να έρχεστε και να μας λέτε τι είναι πολύ σημαντικό για μας και για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ. Maybe, uh, Ίσως αν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Έχουμε μία ετήσια έκδοση ε, δικτών, την παρουσίασα και στο Παρθάν στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι το ίδιο σαν την συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις ημέρες για τον τρόπο με τον οποίο Προσπαθούμε να ε, εντοπίσουμε τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και πώς να ενεργήσουμε στα πλαίσια της νέας πράσινης συμφωνίας. Όλες οι συζητήσεις θα πρέπει να γίνονται με αποδοτικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν μία σειρά δείκτες οι οποίους θα θέλαμε και εμείς και όλοι οι άλλοι να τους λαμβάνουν υπόψη, η Eurostat και άλλες οργανώσεις, ώστε να μπορέσουν να έχει ο κόσμος μία ε, πιο γενική γνώση του τι ακριβώς γίνεται, λαμβάνοντας όλα αυτά τα θέματα υπόψη. Επίσης, τα θέματα που αφορούν τα κονδύλια του προπολογισμού συζητούνται εδώ κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας παρήχε ιδιαίτερος από την δική σας Επιτροπή για τον ε, προϋπολογισμό του 2020 όπου προσθέσαμε προσθέθηκαν κάποιοι πόροι για τον οργανισμό μας και αυτό είναι πρωταρχή σημασία. Γι' αυτό σημαίνει ότι και εμείς χάσαμε πολλά άτομα στο τελευταίο χρόνια λόγω της ε, λιτότητας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι ε, εκτιμώ ιδιαίτερο την προσπάθεια που καταβάλλεται να αυξηθούν τα κονδύλια που μας δόθηκαν. Σας ευχαριστώ. Okay. We are going to resume. Θα συνεχίσουμε τώρα και έχουμε το προνόμιο να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τίμερος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος μετά, λίγες μέρες μετά την παρουσίαση της Πράσινης Συμφωνίας στην Ολομέλεια, μας δίδει την εξαιρετική ευκαιρία να ακούσουμε και περισσότερα από τα γενικά που ακούστηκαν στην Ολομέλεια. Η παρουσίασή του θα διαρκέσει 10-12 λεπτά και μετά θα δώσουμε το λόγο για 2 λεπτά σε κάθε συντονιστή και έχουμε και τον κατάλογο των συναδέλφων. Αρχίζουμε με 10-15 λεπτά για σας κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ. με που είναι εδώ ο και όλα τα άλλα μέλη της ε, αντιπροσωπείας από τη Μαδρίτη. Φτάσατε κιόλας, ε. Για αύριο θα μιλήσουμε στην Ολομέλεια για τη Μαδρίτη, αλλά μπορώ να σας πω σε σχέση με αυτό το θέμα ότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένα τα βλέμματα σε εμά. Το Ευρωπαϊ... Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ε, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στη Μαδρίτη και πολλές φορές προσπάθησα να εξηγήσω περί τίνος πρόκειται διότι η απουσία Αμερικανών ηγετικών στελεχών και η αβεβαιότητα οι Κινέζοι θέλουν και αυτοί να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο ή όχι. Ο ρόλος της Ευρώπης είναι στα πλαίσια της συζήτησης της κλιματικής πρωταρχής σημασίας και βεβαίως ε, θέλουμε να αναλάβουμε εμεί τέτοια ευθύνη, να πρέπει κάτι να προσφέρουμε στον υπόλοιπο κόσμο στα πλαίσια τη Πράσινη Συμφωνία. Για μένα αυτό το οποίο κάνουμε είναι κάτι το οποίο ε, αυτή τη στιγμή από την τελευταία βιομηχανική επανάσταση την οικονομία μας την έχουμε βασίσει στα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε λοιπόν την, ε, να, πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, οικονομία, την ε, ευημερία των πολιτών, την ανάπτυξή μας, να τη βασίσουμε σε κάτι άλλο και όχι στα ορυκτά καύσιμα. Είναι λοιπόν η προσπάθειά μας να αλλάξουμε τα πράγματα και από την οικονομία μας που βασίζεται στον άνθρακα να αποδεσμευτούμε ώστε να μην γίνει, ε, να μην παραμείνει πλέον απειλή επιβίωσης του πλανήτη μας ο άνθρακας. Αυτός λοιπόν είναι κατά την άποψή μου ε, ο κύριος στόχος της Πράσινης Συμφωνίας και βεβαίως πρόκειται για την πιο σημαντικό και προκλητικό αν θέλετε σχέδιο και project Ευρωπαϊκής Ένωσης και μικρή είναι η σύγκριση αν πω τι έγινε με την δημιουργία της ε, ενιαίας αγοράς ή πώς μπόρεσε να δημιουργηθεί η Ευρώπη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πρόκειται για επανεκκίνηση της Ευρώπης και των οικονομιών μας. Βλέπω εδώ συναδέλφους, βλέπω και νέους, οι νέοι μας το ζητούν. Πρέπει κάτι να κάνουμε για τις νεότερες γεγενές. Εμένα Πρόσφατα αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Όσοι είναι σκεπτιστικές ε, για το κλίμα έχουν παιδιά. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς επιβιώνει. Πρέπει να πω ότι ε, τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο από εμά. Και η 16χρονη, την οποία όλοι γνωρίζετε, είναι το πρόσωπο της χρονιάς κατά το Times Magazine και ασχολείται με το κλιματική αλλαγή. Είστε πρωταρχικής σημασίας λοιπόν εσείς ως Επιτροπή, διότι ξεκινάμε από την θεωρία και η δική μας ευθύνη τώρα είναι να το κάνουμε πράξη και νομοθεσία. Τα επόμενα πέντε χρόνια ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε λοιπόν ε, να οδηγήσουμε το όχημα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σε διαφορετική πορεία. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε τον ηγετικό ρόλο και να μπορέσουμε να είμαστε ηγέτες σε θέματα κλιματικά, όπως είπαμε, στα επόμενα, και να είμαστε ουδέτεροι στα επόμενα χρόνια. Ξέρω ότι είναι πολύπλοκο. Μη, ποιες είναι οι αρχές οι οποίες υπογραμμίστηκαν στα πλαίσια ε, της ε, Πράσινης Συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα, ε, τεκμηριωμένα στοιχεία. Νομίζω ότι όταν κάνουμε νομοθετικό έργο εδώ, και το λέω αυτό στα πλαίσια της εμπειρίας μας για την, οδηγίε οδηγίες που αφορούν τα πλαστικά, ότι όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι και καλύτερα επαληθεύσεις τα στοιχεία σου, τόσο πιο καλή νομοθεσία θα κάνεις για να εφαρμοστεί σωστά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε μελέτες αντικτύπου ε, με στάνταρ τρόπο, ώστε να βοηθήσουμε τους συνομοθέτες να εργαστούν καλύτερα για να κάνουν την καλύτερη νομοθεσία. Το επόμενο ε, καλοκαίρι θα γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση ε, του και εκτίμηση τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της κλιματικής ουδετερότητας το 2050. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Η επόμενη ΚΑΠ θα γίνει στη Γλασκόβη και ελπίζω ότι θα μπορέσει να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Αν το κάνουμε αυτό σωστά, στην δική μας ε, αξιολόγηση θα δούμε πώς τους διάφορες τομείς οικονομίας μας, τις ε, μεταφορές, τη γεωργία, την ενέργεια θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και μετά από αυτή την πρώτη εκτίμηση θα αναθεωρήσουμε και θα ε, μεταλλάξουμε όλες τις πολιτικές μας και τους ε, νομοθεσία μας, ώστε να το πλήρες πακέτο να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα τον Ιούνιο του 2021. Δεύτερος πυλώνας. Ποιο είναι το γενικότερο πεδίο εφαρμογή τη Πράσινη Συμφωνία. Το κλίμα. Αλλά το κλίμα σημαίνει επίση ε, περιβάλλον, ε, προστασία της φύσης. Έχουμε ένα οικοσύστημα στο οποίο ζούμε και από το οποίο ζούμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μία διαφορετική φύση στην οποία ζούμε και όχι να συνεχίσουμε επιτιθέμενα στη φύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία αφορά επίση και τη βιοπικιλότητα, δεδομένου ότι χάνονται κάθε χρόνο πολλέ χιλιάδε ε, είδη πανίδε και χλωρίδες. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον μη τοξικό, να έχουμε ασφαλή είδη διατροφής, να κάνουμε σωστή ε, παραγωγή ξυλίας και να έχουμε την ε, βιώσιμη γεωργία και δασοκομεία. Θα θέλουμε βεβαίως να έχουμε πόλεις υγιείς, πράσινες και να, για να το κάνουμε, φτάνω τώρα στον τρίτο πυλώνα, χρειαζόμαστε το μετασχηματισμό της αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στα αυτοκίνητα που οδηγούμε, στα ίδια τροφής που τρώμε, στα σπίτια του ζούμε. Και όλα αυτά βεβαίω σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια νέα βιομηχανική στρατηγική στην Ευρώπη. Και ο τέταρτο πυλώνα είναι τα χρήματα. Τα χρήματα, τα κονδύλια που χρειαζόμαστε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά ε, κονδύλια, επενδύσεις μεγάλες, 250 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να το κάνουμε αυτό το πράγμα διαφορετικά. Το κόστος της ε, μη ενέργειας είναι πολλαπλάσιο. Θα πρέπει λοιπόν <clears throat> να μπορέσουμε να εισαγάγουμε αυτό τον ε, ε, μηχανισμό της δίκαιας μετάβασης και στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το περίφημο Ταμείο της Δίκαιας Μετάφασης. Δεν θα πρέπει να γίνονται παρανομήσεις. Η θα πρέπει η μετάβαση να είναι δίκαια και βεβαίως ξέρουμε ότι μπορούμε να αρχίσουμε με τα κονδύλια, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα μπορέσουμε να δούμε, α, βρούμε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για να μας βοηθήσουν στα πλαίσια αυτού του ταμείου. Και βεβαίως ο τελευταίος σημαντικός και πέμπτος πυλώνας, η συμφωνία η κλιματική. Η πράσινη συμφωνία αφορά τα άτομα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνει από τα άτομα, από τον κόσμο. Θα χρειαζόμαστε τη συμμετοχή του καθενός, των μικρών, των μεγάλων, των νέων, των μεγαλύτερων, από τη, των ε, εργαζομένων, των γεωργών, των ακαδημαϊκών κύκλων, των νέων, των λιγότερων νέων, των πάντων. Το, η συμφωνία λοιπόν αυτή η κλιματική θα πρέπει να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και θα χρειαστώ και τη δική σας σύνδρομη. Όταν θα κάνουμε όλα αυτά σωστά, θα έχουμε κάνει μια εξαιρετική διαδρομή. Και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε σε επανεκκίνηση τις κοινωνίες μας και να δώσουμε ελπίδα στις επόμενες γενιές. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη το να αρχίσει να κάνει ε, αυτή, να, μπει μέσα σε αυτή τη νέα διαδικασία, να ανακαλύψει μια καλύτερη Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι πρόκειται για μια διαδρομή από την οποία δεν υπάρχει γυρισμός. Είναι μονόδρομος και θα πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε ολοκληρώσει για να επιβιώσουμε μέχρι το 2050. Ευχαριστώ. first... Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ε, τα, α, με τους συντονιστές ξεκινάμε τον Πέτερ Λίζα του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πρώτε Αντιπρόεδρε, ξέρετε εκτελεστική Αντιπρόεδρε και συγχαρητήρια για την Πράσινη Συμφωνία. Σε εσά, στην Ursula Φοντερ Λάιν και σε ολόκληρη την Επιτροπή. Εμεί ω ΕΛΚ υποστηρίζουμε πλήρω την πρόταση. Με όλε τι λεπτομέρειε, τη δίκαιη μετάβαση, τη συνεργασία με τη βιομηχανία, τη βιομηχανική στρατηγική και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και που στηρίζεται τόσο την εκτίμηση που Είναι σημαντικό να δούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε πριν πάμε στην νομοθεσία. Να σας συνοψίσω τι συνέβη ε, στη Μαδρίτη. Ήταν απογοητευτικό το τελικό αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία, πάντα λέμε ότι είναι καλύτερο να μην έχει αποτέλεσμα κανένα παρά να έχει κακό αποτέλεσμα. Αλλά δυστυχώ αυτό συνέβη. Στις διμερείς ωστόσο συνεδριάσεις απέκτησα την αίσθηση ότι και πολλές άλλες μεγάλες οικονομίες είναι έτοιμες να συνεργαστούν με την Ευρώπη για μεγαλύτερη φιλοδοξία. Γι' αυτό θα ήθελα να εστιαστώ σε αυτό το κομμάτι της Παρασύνης Συμφωνίας, της επικοινωνίας ε, και της χρήσης όλων των πιθανών εργαλείων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν δράμε μόνοι. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι τα δάση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρομαστε στα δάση. Αλλά όσον αφορά τι συγκεκριμένε δράσει, αναφέρατε ε, ότι πρέπει να φυτευτούν 2 δισεκατομμύρια δέντρα. Από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά από την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά η Κομισιόν πρότεινε να περικοπεί ο δεύτερο πυλώνα. Ενώ αυτό ήταν ο μόνο τρόπο να χρηματοδοτήσουμε τη φύτευση δέντρων για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Και το τελευταίο, δεν ήθελα να σα ενθαρρύνω να συνεχίσετε τη εργασία για την τιμολόγηση του άνθρακα σε μέρη όπου αυτό δεν συμβαίνει ακόμα. Χρειαζόμαστε ένα μείγμα πολιτική, όπω είπατε στην ακρόασή σα. Όχι απλά να δίνουμε εντολέ και να ελέγχουμε, αλλά να έχουμε και μέτρα βασισμένα στην αγορά. Ευχαριστούμε, Γιούτα Γκέτινεν, για του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν. Όπω συνήθω, ε, ε, μα είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από την περασμένη εβδομάδα και την ανακοίνωση της Πράσινης Συμφωνίας ε, και τη συμμετοχή μας στην COP25 ε, αισθάνθηκα περήφανη που είμαι ευρωβουλευτής και που συμμετέχω στα τεκτενόμενα. Ήταν πιο σημαντικό από ό,τι ανέμενα και οι προσδοκίε μου ήταν ήδη μεγάλες, οπότε έχετε μεγάλο φόρτο, μεγάλο βάρος ε, και ε, συμμετείχαμε πολύ καλά στη συζήτηση με τους νέους ανθρώπους ως όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο που αναμένουν από εμάς να φέρουμε αποτελέσματα. Όπω ε, αυτό που κάθεται δίπλα σα, λέει ο κ. Τίμπερμαν. Ναι, μερικέ φορέ ξέρετε η νέα γενιά είναι απαιτητική. Ε, από την Πράσινη Συμφωνία, λοιπόν. Η Πράσινη Συμφωνία θα πετύχει μόνο αν έχουμε με το μέρο μα του πολίτε και αν ε, γίνεται για τους πολίτες και από αυτούς. Ως ε, σοσιαλδημοκράτης λοιπόν και συντονίστρια των σοσιαλδημοκρατών χαίρομαι που αναφέρετε τόσο ε, καθαρά τη δίκαιη μετάβαση και αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Αλλά πάντα φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά. Θα συνεργαστούμε σκληρά μέσα στα επόμενα χρόνια και ιδίω του χρόνου για το ETS. Είναι σαφές πιστεύω ποια είναι η άποψη για τις οδικές μεταφορές εδώ στο Κοινοβούλιο και για το ETS. Θα μπορούσατε να μας αναλύσετε λοιπόν τις ιδέες σας γι' αυτό. Είναι σημαντικό. Επίσης ήθελα να αναφέρω την ναυτιλία. Ξέρω ότι έχετε κάποιες ιδέες για την ναυτιλία και δεν ρωτώ με το 2021 μπορούμε να αναμένουμε να ε, είναι κομμάτι της αναθεώρησης του ETS. Μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό και επίσης ε, θέλετε να δείτε την ε, γραμμική μείωση και ε, την ευθυγράμμιση αυτού με το στόχο του 2030, αλλά αν δείτε και το μερίδιο των ελεύθερων δικαιωμάτων και των ποσών, και αυτό θα ήταν χρήσιμη πληροφορία μετά για τα χημικά. Ξεκινώντα από τη στρατηγική μηδενική ρήπανση, μπορείτε να μα επιβεβαιώσετε ότι ε, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα ε, κατευθύνει τις εργασίες για όλα αυτά, γιατί υπάρχει σύγχυση. Γιατί θέλουμε το περιβάλλον να βρίσκεται στο επίκεντρο της εστίασης. Βλέπετε τόσο πολλά πράγματα γίνονται παγκοσμίω και όσον αφορά την εξαφάνιση ειδών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή πολιτική για τα χημικά επίσης. Ευχαριστούμε. Ρενιού. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε για τον τίτλο σας, γιατί σας παίρνει το μισό χρόνο Όπως γνωρίζετε είμαι 16 χρόνια μεγαλύτερό σας, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω ε, να σας ε, λέμε αγαπητέ Φραντς, στον ενικό. Μετά, μας είπατε να χαράξουμε πορεία. Φυσικά υπάρχουν πολλοί που θέλουν να χαράξουν πορεία και να σχεδιάσουν διάφορα πράγματα. Αν χρειαστεί, λοιπόν, ε, θα πρέπει να βρούμε κάποιον ε, για να χαράξει το χρονοδιάγραμμα. Έρχεται η σύνοδο στην Κίνα, έρχεται η σύνοδο στη Γλασκόβη. Παίρνουμε στα σοβαρά αυτό που συμβαίνει και νομίζω πως πριν την σύνοδο στην Κίνα δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. το επόμενο έτος ε, θα ε, σημάνει το πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για το κλίμα. Θα είναι όντως ένα πλαίσιο και ε, από τι θα αποτελείται αυτό. Θα έχει και στοιχεία για την διακυβέρνηση το 2020, διότι στη δομή της διακυβέρνησης υπάρχουν κάποια σημεία που θέλουν ακόμα επεξεργασία. Μετά, από τη στιγμή που υπάρχει ένα σχέδιο για την δομή αυτής της κλιματικής νομοθεσίας, μετά θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τους νέους στόχους. Το μείον 55% λοιπόν θα πρέπει να ε, ενταχθεί σε αυτούς τους ε, στόχους και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το ποσοστό. Μετά τη Γλασκόβη όλα αυτά. μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες ε, παραπάνω πληροφορίες, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ πρώτα εκτελεστικά την Πρόεδρε Φραντς Τίμερμανς. Εμείς οι Ολλανδοί μια χαρά τα πάμε με τους τίτλους. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την Πράσινη Συμφωνία, διότι επιτέλους κάνουμε στροφή και βάζουμε το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Αν διαβάσετε τις αναλύσεις ε, και τα βασικά σημεία, νομίζω πως ε, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την ε, ανακοίνωση αυτή ως πράσινο μανιφέστο ε, αυτό μπορεί να ανησυχεί κάποιους, ε, όμως ε, φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι η υλοποίηση της νομοθεσίας αυτής, διότι πολλές ανακοινώσεις έχουν γίνει, μας λέτε ότι θα ακολουθήσουν μελέτες, αλλά προκύπτουν και διάφορες συνέπειε και δημιουργούνται ερωτήματα. Καταρχά, σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα, έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι για την βιοπικιλότητα. Υπάρχει απώλεια βιοπικιλότητας που συνεχίζεται. Και φυσικά ένα κομμάτι της ελίσης θα ήταν να, αυξηθούν, να αυξηθεί η έκταση των προστατευόμενων περιοχών, όμως αυτές οι προστατευόμενες περιοχές υφίστανται μεγάλες πιέσεις εξωτερικές. Μετά, η Γεωργία είναι επίση ε, πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια για αλλαγή και φυσικά η μεταρρύθμιση της ε, ΕΚΑΠ που θα ολοκληρωθεί το 2020 θα ε, ισχύει για 7 χρόνια και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα για την νομοθεσία περί βιοπικιλότητας. Δηλαδή πάει λίγο μπροσπίσω πίσω το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς θα το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τι θα κάνουμε με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αν αυτή θα ισχύει μόνο για 7 χρόνια και μετά από 7 χρόνια θα πρέπει να πιάσουμε από την αρχή του νόμου την νομοθεσία για την βιοπικιλότητα. Έπειτα, εμπόριο. Στην Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην εμπορική μας πολιτική. Και με περηφάνεια και καλό σε λέτε ότι μπορούμε πλέον να έχουμε τη Συμφωνία του Παρισιού που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμω στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα έχουμε μια χώρα η οποία υπέγραψε τη Συμφωνία του Παρισιού αλλά δεν την εφαρμόζει και αναφέρομαι στη Βραζιλία και ταυτόχρονα υπάρχει συμφωνία με τη Μερκοσούρ διότι το κεφάλαιο για την ανάπτυξη δεν είναι δεσμευτικό. Γι' αυτό λοιπόν το σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Προτροπή να δει ότι δεν έχει σημασία μόνο η υπογραφή συμφωνιών, αλλά η υλοποίηση. Αυτά είναι τα ουσιώδη που θα κάνουν την διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριο κύριος από το ID. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τίμερμαντς. Δεν αρνούμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε δει τι συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια στο βορρά. Τα πράσινα οικολογικά κόμματα όμως και η ατζέντα τους έχουν θέσει υπερβολικούς τρελούς στόχους που τίποτα κοινό δεν έχουν με την ε, προστασία της άγριας ζωής. Και αυτό το πράσινο όνειρο επιτίθεται στην ε, δασοκομική βιομηχανία της χώρας μου, της Φιλανδίας. Υπάρχουν χώρες με ελάχιστα δέντρα, όμως αυτό δεν συμπεριλαμβάνει και τη Φιλανδία. Αφήστε λοιπόν τα δάση της ε, Φιλανδίας στην ησυχία τους. Ο αυτός ο 1,5 ε, βαθμός είναι η ιερή αγελάδα και συνέχεια επαναλαμβάνεται σαν καραμέλα. Ο ήλιος με τις ακτίνες του δεν έχει καμία ιδέα για αυτόν τον 1,5 βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν ε, εσείς παρουσιάζετε βιβλικές καταστροφές, ε, μας λέτε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου σήμερα. Ε, νομίζω πως υπερβάλλεται και αυτό οδηγεί σε υπερβολές και στην φορολογία και στους στόχους. Αλλά εμείς τι θα πούμε στους πολίτες μας όταν η βενζίνη θα φτάσει τα 3-4 ευρώ το λίτρο. Νομίζω πως είναι ουτοπικό αυτό που λέτε. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι μεγαλύτερες από ό,τι ε, τον δίζελ, αν δούμε όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Γιατί λοιπόν ε, η συμφωνία του Παρισιού έδωσε το ελεύθερο στην Κίνα να ρηπαίνει. Και εμείς έχουμε βάλει ίδια τη θηλιά στο λαιμό μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάτι να γίνει. Όλοι έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας και κάθε εποχή έχει και τις παραξενιές της και αυτή η παράνοια για το κλίμα είναι η τρέλα της εποχής. Όμως ε, νομίζω πως χρειάζεται λίγη κοινή λογική εδώ. Μάλιστα ο Αλεξάντερ Βόντρα από την ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλή τύχη. Είστε ένα από τα λαμπρότερα μυαλά και ένας από τους καλύτερους ε, επιτρόπους ε, σε θέματα επικοινωνίας που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μιλάμε για μια επανάσταση. Η επανάσταση είναι μια λέξη που μπορούμε εύκολα να πουλήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, δύσκολα όμως στους Ευρωπαίους πολίτες. Ιδιαίτερα μάλιστα αν αναλογιστεί κάποιο και τις συνέπειες που έχει αυτή η επανάσταση. Χρειαζόμαστε αξιόπιστους και εφικτούς κλιματικούς στόχους, όμως ε, οι στόχοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ε, από ό,τι βλέπω στο κείμενο, μας προκαλούν ανησυχίες. Μας προκαλούν ανησυχίες επίσης και οι διαδικασίες που προβλέπονται και η χρηματοδότηση που προβλέπεται, αλλά και οι πιθανές εντάσεις που αυτή η νομοθεσία θα δημιουργήσει εντός της Ευρώπης αλλά και εκτός της. Τώρα, ως προς την ε, διαδικασία. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και σε ό,τι φορά την φιλοδοξία, να σας πω ότι πριν από μια ώρα είχαμε εδώ συζήτηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ετήσια έκθεση και μιλάγαμε για τους στόχους του 2020. Επτά από 27 τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται ε, στα όρια, έχουν οριακές τιμές ε, σε ό,τι αφορά αυτού τους στόχους. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα αξιοπιστίας. Μετά, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση αυτού του οράματος, του κοινού οράματος, της κοινή στρατηγικής, δηλαδή της ε, δημιουργίας πόρων και δεδομένων και των εντάσεων εντός και εκτός Ευρώπης, νομίζω πως δημιουργεί δυσκολίες. Ε, το είπε και ο Μάρεκ. Και μάλιστα αυτές οι δυσκολίες είναι αισθητέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η καγκελάριος Μέρκελ το είπε ότι αυτή η προσαρμογή του άνθρακα θα οδηγήσει σε εμπορικό οικονομικό πόλεμο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την Γκουέ Σισιαμονίκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμαντς, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε απόψε για να συζητήσετε μαζί μας αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και το πολύ σημαντικό μήνυμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή αν ασχοληθούμε σφαιρικά. Αυτή η δίκαιη μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιοι σε όλους τους τομείς επίσης και πρέπει να συνεργαστούν όλοι και ο γεωργικός τομέας και οι μεταφορές και η επισητιστική βιομηχανία αλλά κυρίως οι πολίτες. Και για τους σοσιαλιστές είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, αυτή η διάσταση. Όμως με ανησυχεί το ότι για να είμαστε ε, ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα, όπως είχαμε πει το 2015, θα πρέπει να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους. Ο στόχος ε, του 30% μέχρι το 2030 ήταν αρκετά φιλόδοξος από μόνος του. Τώρα μας λέτε για 55% μέχρι το 2050, αλλά το 55% είναι η ελάχιστη τιμή που πρέπει να πιάσουμε. Και δεδομένου μάλιστα, δεδομένων μάλιστα των εξελίξεων ε, είναι προφανές ότι εάν οι στόχοι δεν είναι επαρκείς, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με μία άνευ προηγουμένου κατάσταση που θα πρέπει να μας κάνει να αλλάξουμε 180 μοίρες στο σκεπτικό μας. Και να ξέρετε ότι εάν φτάσουμε στο προχώρητο θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πώς λοιπόν θα συμπεριληφθούν όλα αυτά στη μελλοντική νομοθεσία. Εάν δεν έχει αποτέλεσμα η δέσμευση του άνθρακα, τι θα γίνει στον ε, γεωργικό κλάδο. Σίγουρα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Αλλά εσείς πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι και ο γεωργικός κλάδος θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Όμως ε, επαναλαμβάνω ότι αν δεν αλλάξουμε ε, τον ε, τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη γεωργία δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Και στην Φιλανδία, κυρία Χακαλάινεν. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τη βιοπικιλότητα ούτε στη Φιλανδία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας στη βιοενέργεια από τα δάση. Πρέπει να δούμε πώς ε, λειτουργούν αυτοί οι αποθετήρες άνθρακα και να αναπροσαρμόσουμε την ε, δασική μας στρατηγική. Ευχαριστώ. Για 10 λεπτά έχετε το λόγο. σωστά είπε αυτά τα οποία ο κύριος Λίζε. Θα έχουμε ένα τρομερό καθήκον τα επόμενα χρόνια. Με, να αναπτύξουμε ε, μία νέα διπλωματία με άλλα κράτη. Καλό και κακό αυτό. Κλιματική δημοκρατία. Όταν το παρουσίασα είπα κάτι το οποίο ενδιέφερε ε, πάρα πολύ κόσμο, τη Χιλή, την Κολομβία, άλλου. Πώ θα το κάνετε. Αυτό έγινε μετά την προσήλωση του Green Deal. Βεβαίω, υπάρχουν άλλοι μεγάλοι παίκτες. Η Κίνα που είναι ακόμη σε αμυντική θέση. Περιμένει να δει, να κάνουμε, να δείξουμε εμεί τι κάνουμε, να έρθουμε σε επαφή. Η Βραζιλία μπλοκάρει σαφώ τα πράγματα και δημιουργεί συμμαχίε με χώρε που ήταν πολύ πιο κοντινέ παλιά με μας, τι Αφρικανικέ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την διπλωματία μας με χώρες της Αφρικής που είναι επί της ε, ουσίας σύμφωνοι και πιστεύουμε ότι άλλοι τους έχουν εγκαταλείψει. Σωστά λοιπόν είπατε ότι πραγματικά χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη διπλωματία σε θέματα κλιματικά και Μπορείτε να πεις, Μανφρέτ, ότι το έχω, το έχω. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Για τα δάση. Επίσης, σωστά είπες ότι θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι έχουμε τα κατάλληλα κονδύλια. Βεβαίω θα πρέπει να κινητοποιηθούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και διαρωτώ με για τον, στον πρώτο πυλώνα, θα το μελετήσουμε αυτό, και ο πρώτος πυλώνας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από ό,τι τώρα στην ε, να δούμε προς τα που πάμε, αλλά θα πρέπει ακόμη τους επόμενους μήνες να το συζητήσουμε. Επίσης, για τα, μέτρα μας, για τα δάση. Είναι φτηνότερα από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και είναι επίσης μια ευκαιρία και για την ε, γεωργία και για την βελτίωση των πόλεων, να τις κάνουμε πιο πράσινες, να βοηθήσουμε ό, την ε, ποικιλότητα. Είναι πολύ λίγα τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται για την ε, ε, επαναδάσωση της Ευρώπης. Αλλά και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πει σε κάποιον ε, και πολύ πιο απλό ότι πρέπει να φυτέψεις δέντρα και να κάνεις νέα δάση παρά να μιλάς για άλλα θέματα, για το ίστιες. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε με ευφύ τρόπο. Το να προσπαθήσει κανείς να ε, φυτέψει δέντρα σε άγωνα δεν είναι έξυπνο, αλλά το να προσπαθήσουμε εκεί που έχουν γίνει κάποιες αποψηλώσεις, να ξαναβοηθήσουμε τα δάση να αναγεννηθούν είναι εύκολο. Και πάλι συμφωνώ μαζί σου, θα στο έξω, συνέχεια συμφωνώ μαζί σου, αλλά εν Απόψε είναι μια ειδική ημέρα. Ε, τώρα, εάν έμαθα κάτι στη Μαδρίτη, είναι ότι πραγματικά όταν αυξάνεται η τιμή του άνθρακα, οι κάποιες πηγές, ενέργειας δεν είναι πλέον βιώσιμες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να, ε, να εγκαταλείψουμε τον άνθρακα. Επίσης, ε, η στα θέματα των ναυτιλιακών μεταφορών. Θα πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, ας το θέσουμε ε, ως εξής. Θα πρέπει να έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία για να δούμε τι κάνουμε. Αλλά ας το δούμε, ας το διαβάσουμε. Χαίρομαι αν με πείσει κάποιος ότι αυτή είναι καλή ιδέα, αλλά αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι πεπισμένοι. Επίσης, αν αποδειχθεί ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως πιστεύουν, θα πρέπει και εκείνοι να αλλάξουν δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα επιλέξουμε σε αυτό το Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί σε θέματα των ε, ε, ελευθέρων ποσοτήτων ε, ή των μέτρων που δίδονται, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το χειριστούμε αυτό πιο, με πιο αυστηρούς κανόνες. Στρατηγική μηδενικής ρήπανσης. Ποια είναι η γενική διεύθυνση που ηγείται όλες αυτές τις πολιτικές. Η ένβη, αναμφίβολα. Διότι πιστεύω ειλικρινά ή για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες, για τα χημικά προϊόντα, για τα φυτοφάρμακα. Πιστεύω ειλικρινά ότι η επίθεση όλων αυτών των στοιχείων ε, συνδυασμένων στον άνθρωπο είναι πραγματικά μεγάλη και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Τώρα, χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, Νίλ. αυτό είναι το θέμα. Εάν αρχίσεις λέγοντας θέλουμε να είμαστε το 2050 κλιματικά ουδέτεροι, δεν έχεις καμία επιλογή. Αλλά ας δούμε από το 20 πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλη την πολιτική μας ώστε να καταλήξουμε έτσι Και βεβαίως αυτό θα έχει και διάφορες επιπτώσεις στην σχετική νομοθεσία περί κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να το δούμε από πάρα πολλές οπτικές γωνίες. Yeah. Yeah. This is not a language I speak. I used to. Δεν μιλάω πια αυτή τη γλώσσα. Την μιλούσα όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, αλλά τώρα πάει. Την ξέχασα. Και θα σας πω το εξής. στη σχετική νομοθεσία για το κλίμα θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και ακριβείς για να δούμε ε, σε λεπτομέρειες τι θα κάνουμε. Ε, κάτι χρήσιμο, όχι να πούμε απλώς πρέπει να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι μέχρι το 50, παύλα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με μεγάλη ακρίβεια από νομικής πλευράς, και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τρόπο που να μην μιλάμε για το τέλος το 2050, αλλά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε προοδευτικά, 20, 30 κτλ. Και η νομοθεσία σχετική δεν θα πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής ή εάν δούμε ότι αυτό είναι χρήσιμο. Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια, ό,τι αφορούσε την, πέντε χρόνια πριν, την ηλιακή ενέργεια, την αιωλική, δεν ξέραμε πράγματα που τα ξέρουμε σήμερα και αν δεν είχαμε επιτρέψει να γίνονται αλλαγές, πού θα πηγαίναμε. Διότι πιστεύω γενικά ότι από τότε ότι η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια είναι διαφορετικές από τα καύσιμα, ε, θα πρέπει να δείτε πού μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην αποθήκευση και στην ε, διανομή ίσως να υπάρχει πρόβλημα. Σας το λέω αυτό ως παράδειγμα. Άρα θα πρέπει κανείς να μπορεί να αλλάξει τα πράγματα αν δει ότι κάτι δεν πάει κολλά. Και βεβαίως ο σχεδιασμός της ε, επόμενης ε, ε διάσκεψη τη βιοπικιλότητα του χρόνου στην ε, Κίνα είναι κάτι το δύσκολο, διότι δεν έχουμε βάση από την οποία να ξεκινήσουμε. Κάτι το συγκεκριμένο δηλαδή. Προσπαθούμε λοιπόν στις υπηρεσίες μας να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από το οποίο να ξεκινήσουμε. Όσον αφορά τώρα τι εμπορικέ συμφωνίε, εάν πούμε ότι θέλουμε να είναι δεσμευτικές, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις παρούσες συμφωνίε. και εάν όχι ε, να, να κάνουμε ευθύ εξ αρχή απαγόρευση, να κάνουμε σχεδόν απαγόρευση. Δηλαδή, να πούμε στους πολίτες μας ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ότι τα πρότυπα που ακολουθούμε δεν θα μας οδηγήσουν σε αποψήλωση των δασών. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε σχεδόν δεσμευτικές ε, συμφωνίες με τις χώρες Μερκοσούρ. Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ειλικρινά πιστεύω ότι εάν δεν αλλάξουμε τις βασικές παραμέτρους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και διαρωτώ διαρωτώ με κατά πόσο θα πρέπει να αποδειχθούμε πιο δημιουργικοί και για το δεύτερο πυλώνα, αλλά και για τα επιπλέον πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Θέλω να το δούμε το επόμενο δίμηνο αυτό με τους συναδέλφους μου ε, που ασχολούνται με τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο που θα σας παρουσιάσουν την Άνοιξη και θα σας ακουστώ λίγο εικονοπλάστης τώρα αλλά αν πάτε να δείτε την τελευταία 20 αιτία τι ακριβώς μορφή είχε η ΚΑΠ. Λέγαμε στους αγρότες, εντάξει, μην μιλάτε και πολύ και μην διαμαρτύρεστε και πολύ, να σας δώσουμε κάποια λεφτά και τέλος. Είστε ένα μικρό κομμάτι της οικονομίας μας, να έχουμε ιστορία ως Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε κάτι για εσάς κτλ. κτλ. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε την προσέγγιση και την πρόταση προς αυτούς. Χρειαζόμαστε περισσότερη γεωργία και όχι λιγότερη στο μέλλον, αλλά πρέπει να γίνεται διαφορετικά, ούτως ώστε η γεωργία αυτή να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσει για τα ζυζανιοκτώνα, για τη βιοπικιλότητα, για την προστασία γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, μια νέα συμφωνία που θα συνάψουμε με την γεωργική κοινότητα. Τους χρειαζόμαστε τους γεωργούς περισσότερο από παλιά. Από την πολιτική μου οικογένεια αυτό δεν ακούγεται καθημερινά, ίσως, αλλά εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Με λυπεί να βλέπω γεωργούς να κατεβαίνουν στους δρόμους για να προσπαθήσουν να προστατεύσουν το σύστημα που δεν τους διασφαλίζει μέλλον. Αυτό είναι το λυπηρό. Και στη χώρα μου ακόμα κατεβαίνουν στους δρόμους επιθετικά οι γεωργοί υπερασπιζόμενοι ένα σύστημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα τους προσφέρει ένα μέλλον. Εγώ θέλω να σταθώ δίπλα σε αυτούς ε, τους γεωργούς, να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα που θα έχει μέλλον και ελπίζω και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο η Επιτροπή Άγκρε αλλά και η δική σας Επιτροπή να συμμετέχει στον επανασχεδιασμό αυτού του συστήματος. Το υπερασπίζω στεναρά, γιατί αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα των ανθρώπων που κατεβαίνουν στους δρόμους φυσικά. Τώρα, ε, η τρέλα και το κλίμα που είπατε. Να σας πω ένα πράγμα. Οι πιο πολλοί από εμάς εδώ είμαστε παιδιά του διαφωτισμού και τα παιδιά του διαφωτισμού έχουν αυτό το παράξενο χαρακτηριστικό ότι αφήνονται να τους καθοδηγούν τα δεδομένα, τα στοιχεία και οι επιστήμες. Μέχρι στιγμής η επιστήμη, τα επιστημονικά στοιχεία είναι διαφυσβήτητα θα έλεγα και το λέω απλά και ηρεμά. Είναι μάλλον αδιαφυσβήτητα. Και θα ήταν όχι μόνο πολιτικό αλλά και ηθικό έγκλημα το να τα ξέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να μην κάνουμε τίποτα. Είναι ανάγκη, δεν είναι πια πολυτέλεια, ούτε απλά μια ευκαιρία. Είναι μια ανάγκη. Αν ξαφνικά ανακαλύπταμε ένα κομίτι σε 30 χρόνια που έρχεται προς τη γη, θα λέγαμε «Α, ιστερία, ας ε, στρέψουμε τα μάτια μας αλλού». Όχι, θα κάναμε ό,τι προσπάθεια ήταν δυνατό για να αποφύγουμε την καταστροφή. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τώρα. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε ως ανθρωπότητα για να αποτρέψουμε την καταστροφή αυτή. Για το μηχανισμό προσαρμογής ε, στα σύνορα, για τον άνθρακα. Να σας πω, προερχόμενος, ε, καθώς μόλις ήρθα από τη Μαδρίτη, αν οι χώρες που συνυπέγραψαν το Παρίσι δεν αναλάβουν μέτρα για να εφαρμόσουν το Παρίσι, η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι για να υλοποιηθεί το Παρίσι δεν μπορώ να στραφώ και να λέω στη βιομηχανία μα και στην οικονομία μα πρέπει να κάνετε τεράστιε επενδύσει για να απαλλαγείτε από τι ανθρακούχε εκπομπέ και ξαφνικά να έχουμε τεράστιε διαρροέ που θα σκοτώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Απαράδεκτο. Ίσως το λαδικό μου DNA μου λέει ότι δεν μου αρέσουν εμπορικοί πόλεμοι ούτε εμπορικοί φραγμοί. Καθόλου. Αλλά αν χρειαστεί να ε, κάνουμε κάτι τέτοιο κάποια χρόνια ε, θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα. Ε, δεν είναι, να μην είναι, χρειαστεί η προσαρμογή στα σύνορα, θα πηγαίνει. Μπορεί να γίνει ως φόρο στα σύνορα ε, επιπροϊόντων, ε, ο καθορισμός του ανθρακικού αποτύπωματος κάποιων προϊόντων και προσαρμογή του μηχανισμού μέσω του συστήματος ETS. Επίσης θα μπορούσαν να βρεθούν τρόποι. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό. Απάντησα νομίζω σε όλες τις ερωτήσεις και για τη Γεωργία απάντησα ήδη και για τα δάση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων και ξεκινάμε ε, με την Εστεντελάνγκη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με φέρετε σε δύσκολη θέση εδώ. Εγώ θα μιλούσα για την πράσινη διπλωματία και τα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα εκεί. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Οι γεωργοί που κατεβαίνουν στους δρόμους στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις κάτω Πρώτα απ' όλα θέλουν κάποια αναγνώριση. Και μετά τον έρχεται κανείς και να λέει ότι η ΚΑΠ ουσιαστικά δεν είναι για σας τόσο πολύ, δεν είστε τόσο σημαντικοί, είστε μικρός τομέας, απλά βουλώστε το. Ε, είναι το τελευταίο που χρειάζεται να ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε εγώ ανησυχώ με αυτό που προτείνεται και πρέπει να το πω καθαρά. Ε, κατά κάποιο τρόπο έτσι είπε. Τώρα να τους που λέμε μη μιλάτε και δεν είστε σημαντικοί. Δεν, αυτό είπατε, αλλά θέλω να... Ε, ε, είμαι αισιόδοξη και να πω κάτι θετικό που είπατε εδώ πέρα. Είπατε δημιουργική σκέψη. Να πάρουμε περισσότερα χρήματα από τον πρώτο πυλώνα, να σκεφτούμε ε, θετικά και δημιουργικά για να δούμε πώς θα είναι η μελλοντική ΚΑΠ. αυτό είναι θετικό. Αλλά μιλήστε και για κρατικές ενισχύσεις. Για να σκεφτούμε δημιουργικά χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι όταν δίνουμε 74 σέντ το κιλό για τα λαχανά και Βρυξελών στον αγρότη, για 90, τόσο λίγο δηλαδή, ε, κάτω από το μισό δίνουμε στον αγρότη από τα προϊόντα που αγοράζουμε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Υπάρχει τεράστια διαφορά από τα πόσα πληρώνουμε και πόσα λαμβάνουν αυτοί. Οπότε οι κρατικοί κανόνε, ε, οι κανόνε κρατική ενίσχυση θα μπορούσαν να βοηθήσουν να του πούμε ότι κάνετε περισσότερα για τη βιοπικιλότητα το οποίο σημαίνει ότι η παραγωγή σας ε, κοστίζει περισσότερο, οπότε ας επιτρέψουμε να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες επιτιμών σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο όφελος για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Οπότε η ερώτησή μου προς τον κύριο Τίμερμαντζ είναι πώς θα πείσετε την Αντιπρόεδρο Φεστάγκερ να σκεφτεί δημιουργικά βάσει όλων αυτών, γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια λύση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρατηρείτε το ένα λεπτό, αν θέλετε. Ε, σοσιαλιστές. Καλά που το λέτε την ώρα που πήρα εγώ το μικρόφωνο. Λοιπόν, κύριε πρώτη αντιπρόεδρε, κύριε ε, Φραντς, αγαπητέ Φράνς να σας συγχαρώ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα συνδυασμού κλιματικής δικαιοσύνης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό. Τα δύο αυτά πρέπει να να πηγαίνουν μαζί είναι καταπληκτικό βήμα ώστε η Ευρώπη να μειώσει τις ε, εκπομπές και να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2050. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει τα περισσότερα αγαθά στον κόσμο με αυξανόμενο ανθρακικό αποτύπωμα, αν σκεφτεί κανεί ε, την κατανάλωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι εισάγουμε πολλά καταναλωτικά προϊόντα από χώρε εκτό Ευρώπη για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή και τη δημιουργία ενό βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη μας χρειάζεται να μετριάσουμε τις εκπομπές μας και ο μηχανισμός ε, προσαρμογής στα σύνορα μπορεί να είναι ένας τρόπος να αποτελέσει κίνητρο για παραγωγούς εκτός ευρωπαϊκής αγοράς να παράγουν πιο βιώσιμα και η ερώτησή μου είναι υπάρχει και αναλλακτική λύση για αυτό το μηχανισμό προσαρμογής στα σύνορα ε, πρότυπα βιωσιμότητας για τα προϊόντα και τα ε, ημιτελή προϊόντα. Θα μπορούσε να είναι μία απέτηση έντασης άνθρακα για προϊόντα όπως ο χάλιβας, όπως είπατε, και να επεκτείνουμε τις απαιτήσει οικολογικού σχεδιασμού να συμπεριλαμβάνουν και τα πρώτε ύλε και τα ημιτελή προϊόντα. Ε, με περίεργο να ακούσω τι έχετε να πείτε για αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Ροντρίγκης Ραμός από το Ρινιού. No. Yeah. Ε, Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Μόλις φτάσετε από τη Μαδρίτη. Είναι αλήθεια ότι είναι αναμφισβήτητη σε αυτή τη ε, διάσκεψη ο ηγετικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποια απογοητευτικά αποτελέσματα. Μεγάλες χώρες που ρηπαίνουν, οι οποίες αρνούνται εφόσον υπέγραψαν, εφαρμόσουν αυτά που υπέγραψαν. Και ο καλύτερο τρόπος για να προχωρήσουν τα πράγματα είναι να προχωρήσουμε εμείς περισσότερο. Αν δεν θέλουν να προχωρήσουν στο άρθρο 6, θα πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα στα οποία κατά κάποιο τρόπο να υποχρεώνονται να αγοράζουν τις ποσοστώσεις άνθρακα. Θα πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό. Αλλά μία καινοτόμος μη ρηπογόνος ευρωπαϊκή ε, επιχείρηση θα πρέπει να προστατεύεται. Επίσης, πιστεύω ότι η... η ετικέτα στα διάφορα προϊόντα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής να ξέρει ο κάθε καταναλωτής τι αγοράζει. Επίσης, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε κανένα στόχο της βιοπικιλότητας εάν δεν υπολογίζουμε στους αγρότες. Και τώρα πρέπει να τους πούμε με ειλικρίνεια, πραγματικά σας χρειάζεται η Ευρώπη με μια διαφορετική γεωργία. Σας ευχαριστώ για το ΕΛΚ και πάλι εντυνάτελση. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Χαιρετίζω την Ευρωπαϊκή Συμφωνία που είναι η πρώτη ευρωπαϊκή συμφωνία για να σωθεί ο πλανήτης μας. Και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δοθούν τα κατάλληλα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην υπάρχει συμπληρωματικό κόστος για τους ε, καταναλωτές. Το να αυξηθεί η τιμή των τροφίμων δεν μπορεί να γίνει αποδεικτό. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις που να σέβονται τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και να βοηθήσουμε και τις πιο μακρισμένες και φτωχές περιοχές της Ευρώπης. Η πράσινη λοιπόν συμφωνία δεν θα πρέπει να είναι μόνο φιλόδοξη, να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών και να προστατεύει τους καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μου είναι πώς θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι καμία πόλη, καμία περιοχή και κανένα άτομο δεν θα ε, μπει στο περιθώριο στα πλαίσια αυτής της μετάβασης και τι ακριβώς θα γίνει με τα κονδύλια που θα δοθούν σε αυτό τον μηχανισμό της δίκαιας μετάβασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για την COP25 και για τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Βεβαίως, ο ιδιωτικός ρόλος που μπορούμε να παίξουμε ως Ευρώπη είναι προφανή. Η πράσινη συμφωνία δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε και νομιμότητα σε σχέση με τους πολίτες μας και να μπορέσουμε σε όλο τον κόσμο να προασπίσουμε τις ιδέες μας και όσοι θέλουν να βάλουν σύνορα για να μην γίνουν αλλαγές, δεν μπορούν να το κάνουν. Τώρα, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να μην μποϊκοτάρουμε τίποτε το θετικό. Θα θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Συμβαίνει κάπως κάτι στο Συμβούλιο. Θα ήθελε κύριε Αντιπρόεδρε να μου πείτε, μήπως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι κάπως ε, ατελή για το στόχους μας. Μήπως αυτό μπορεί να αποτελέσει κάτι το αρνητικό για την υλοποίηση της ε, πράσινης συμφωνίας. Ήταν θετικά τα συμπερασματά τους, αλλά όχι και ομόφωνα τώρα. Όσον αφορά το Ταμείο της Δίκαιας Μετάβασης, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές θα πρέπει να ξέρουμε όμως πού θα βρεθούν τα κονδύλια. Πού θα Πώς θα μπορέσουμε να ε, βρούμε κονδύλια από τα διάφορα ταμεία, θα, κάνουμε, θα έχουμε και ειδικού πόρους εκεί, τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει να το δούμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να επανέλθω στην στρατηγική από το, από το χωράφι στο πιάτο μας. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να ε, μειώσουμε την κλιματική αλλαγή, δεν έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάτε ε, αυτές τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε, ότι τις έχετε κάνει σε όλους τους τομείς. Τι θα κάνετε με το θέμα της ε, κτηνοτροφίας. Υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά θέματα και τα διάφορα ε, εδάφη που χρησιμοποιούνται πραγματικά είναι σε κακή κατάσταση. Άρα, απ' την άλλη, θέλουμε να εισάγουμε τα προϊόντα που δεν έχουμε. Άρα δεν είναι βιώσιμα όλα αυτά. Πότε λοιπόν θα έχουμε μια στρατηγική που θα κάνει αξιοποίηση των οικολογικών αντικτύπων των ειδών διατροφής μας και πότε θα μπορέσουμε να συνάγουμε τα, ε, στα συμπεράσματα. Πότε θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις στην εντατική κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Η Ζωέλ Μελό συνεχίζει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχετε στα χέρια σας ένα οδικό χάρτη που ορισμένοι επαγγελματίες του μάρκετινγκ στην Κομισιόν ονόμασαν Green New Deal, νέα πράσινη συμφωνία. Αν θεωρήσουμε ότι το κλίμα, το περιβάλλον, η βιοπικιλότητα, η ωκεανή, ο αέρας ε, και το τοπίο βρίσκονται σε κίνδυνο, αυτό είναι γιατί μεταξύ άλλων οι, όσοι λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν σε ένα τεράστιο οικονομικό έργο στις τέσσερις γωνιές της γης. Και σήμερα μπροστά στην αποτυχία των παλιότερων σας πολιτικών προσπαθείτε να βάψετε πράσινες όλες τις νέες στρατηγικές σας για την ανάπτυξη στην Ευρώπη και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ευρωπαϊκά του. Υποστηρίζετε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών, ενώ θα έπρεπε να υποστηρίζετε καινοτομία στα πυρηνικά, δεν το συζητάτε. Και εκεί που θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Γεωργία να βρίσκεται στην πρώτη θέση, εσεί την παρατάτε στα χέρια της, του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Απόψε έχετε την ευκαιρία να δώσετε ελπίδα στου Ευρωπαίου. Μπορείτε μπροστά μα να δεσμευτείτε να δώσουμε τέλο στι ε, συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών που είναι μη οικολογικέ και που υπονομεύουν ε, την παραγωγή που υπάρχει στην Ευρώπη, μετατοπίζοντάς τη σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Πάμε στον τελευταίο γύρο και μετά θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Οι τελευταίοι επτά ομιλητές στα Νισλάφ ε, Πολτσάκ για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιμερμάνς, για τη θετική σας τάση. Και νομίζω πως η συνέχεια που έχετε δώσει στις ανακοινώσεις της Φοντερ Λάιν είναι ε, πάρα πολύ καλή. Ε, έχω μια ερώτηση σχετικά με την ε, δασοκομεία. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο οικονομικές πτυχές, αλλά οι αρμοδιότητες. Τα δάση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη έκταση ε, στον πλανήτη μας. Κάτι που μόλις ε, μας είπε ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Χρειάζεται λοιπόν οργανωμένη δράση για την διαχείριση των δασών. Ποια λοιπόν είναι η προσέγγιση που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ρόλο θα διαδραματίσουν τα κράτη-μέλη. Διότι η διαχείριση των δασών σίγουρα πρέπει να αλλάξει. Αυτό έχουν ε, πει σχεδόν όλοι. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό και ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες που θα μείνουν στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Στανιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συνεδρίαση ήταν όντως ε, μη αναμενόμενη. Ήταν ε, να έχουμε διαφορετική ε, τροπή στη συζήτηση. Σε λίγες ε, μέρες λοιπόν ε, θα έχουμε την τελική πρόταση για το κλίμα. Αναφέρθηκε επίση το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για το κλίμα. Θα μπορούσατε να γίνετε πιο συγκεκριμένο πώ θα δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια, πώ θα γίνει η χρηματοδότηση τα ερχόμενα έτη. Και πώς ακριβώς θα συμβάλλουν σε αυτήν την μετάβαση. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας ε, δώσετε περισσότερα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, γιατί μας είπατε ότι μένουν 80 μέρες πριν την ε, παρουσίαση της ε, νομοθεσίας, αλλά από την άλλη έχουμε και την συμφωνία του Παρισιού με τις Ηνωμένε Πολιτείες να αποχωρούν και μετά ακούμε διάφορες αντίθετες μεταξύ τους απόψεις και εγώ προσωπικά νομίζω πως ε, το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο για αυτή τη μετάβαση. Είμαι από την Πολωνία, ένα από τα κράτη που έπεσαν θύματα του κομμουνιστικού καθεστώτος, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όλο, και υπέστη η χώρα μου όλους, ε, όλες αυτές ε, τις αλλαγές. Και ο λαό τη Πολωνία απέδειξε με τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι σε θέση να επενδύσει και να κάνει αυτήν την ε, ιδέα πραγματικότητα. Γι' αυτό νομίζω πως ε, του οφείλουμε λίγο σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ για το Ρηνιού, κυρία Στεφανότα. Κύριε Στεφανότα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τίμερμαντς, δεν ξέρω αν σας προσφώνησε κανεί έτσι. Έχω δύο ερωτήσει. Πρώτον, η μη εφαρμογή και η μη συμμόρφωση. Ήδη έχουμε αρκετά καλή νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να δημιουργείται η εντύπωση ότι η Πράσινη Συμφωνία έχει να κάνει με νέες ε, ιδέες και νέες προτάσεις. Έχει να κάνει και με την ε, εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Υπάρχουν κράτη-μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία επί γιατί δεν συμμορφώνονται. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες δεν πιάνουν τα όρια και αναγκάζονται να πληρώσουν πρόστιμα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και πολιτικά και αλλιώ. Έπειτα, αποψήλωση των δασών. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεστε στο θέμα. Στη χώρα μου έχουμε 3 ε, έως 9 εκτάρια δασικής έκτασης που χάνονται από την παράτομη, παράνομη υλοτομία κάθε χρόνο. Όπως είπε και ο Νέβιλ Τσάμπερλεν ε, δεν πρόκειται για ένα μακρινό μέρος που κανείς δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό. Όχι. Η αποψήλωση των δασών συμβαίνει εδώ στην επικράτειά μας, εδώ στα σπίτια μας. Γι' αυτό και ω συνέχεια της πρότασης του κύριου Λίζε θα σας ρωτούσα ποια είναι η αποψή σας ε, για το ξεκίνημα ενός νέου project που θα στο οποίο θα συμμετάσχουν και νέοι, δηλαδή κάποια κουπόνια για αναδάσωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος, ε, κύριε Μπουρκάρτ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτής της πολύ καλής πράσινης ε, συμφωνίας. Να διαφωνήσω με τον πλησίδη. Εγώ συμφωνώ ότι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή για το κλίμα και για τους πολίτες. Και νομίζω πως από την συζήτηση που γίνεται εδώ καταλαβαίνουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θέλει να γίνει συζήτηση, να γίνει διάλογος έτσι ώστε να ε, παγιοποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Είναι πολύ καλό λοιπόν που ήρθατε εδώ και παρουσιάζετε αυτή την πράσινη συμφωνία. Είναι μια νέα επιτροπή με μια νέα φρέσκια πρόταση. Ήδη ακούσαμε τον Ιούλιο τον πρόδρομο αυτής ε, της πρότασης με τις με τα ποσοστά, με τις αλλαγές ε, που γίνονται και τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά που έχουν οδηγήσει στην ε, επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Νομίζω όμως ότι τα εθελοντικά μέτρα και οι διάφορες ταμπέλες δεν θα βοηθήσουν πουθενά. Χρειάζεται να δούμε ότι ο καταναλωτής δεν είναι χαζός, ότι καταλαβαίνει όταν πρόκειται για πράσινο ξέπλυμα. Χρειάζεται να δούμε όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Χρειάζεται να δούμε ο ποιος είναι υπεύθυνος. Χρειάζεται επίσης να αναγνωρίσουμε ότι πολλές φορές ε, μεταθέτουμε τις ευθύνες μας στα κράτη-μέλη και από, στα σε τρίτα κράτη και τα τρίτα κράτη μετά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ευχαριστώ ε, πολύ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, αναφερθήκατε στη νέα στρατηγική για τα δάση. Θα μπορούσατε να μας ε, πείτε στη νέα στρατηγική ποιος είναι ο λόγος αποψήλωσης με αναδάσωσης. Δεν ε, λαμβάνονται πολλά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την απώλεια της βιοπικιλότητας και βλέπουμε ότι χάνονται πολλά εκτάρια δάσους κάθε χρόνο και οι προσπάθειες για αναδάσωση όμως ε, δεν υπολογίζουν την ε, ήδη υπάρχουσα χλωρίδα. Έχουμε κονοφόρα δέντρα τα οποία δεν είναι ενδυμικά σε περιοχές όπου γίνεται αναδάσωση. Επίσης, η βιομάζα θεωρείται ουδέτερη ως προς το αποτύπωμα άνθρακα. Εσείς ε, τι γνώμη έχετε γι' αυτά και επίσης ε, πιστεύετε πως η βιομάζα δεν είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα. Η Πράσινη Συμφωνία δεν παρακίνησε και άλλες χώρες στην ανάληψη δράσης, έτσι όπως ελπίζατε. Τι θεωρείτε πως πρέπει να γίνει για να βγούμε από αυτό το πολιτικό διέξοδο... έτσι ώστε η COP26 στην Γλασκόβη να είναι πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Εύη για τους μη αναγεγραμμένους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στον ε, μηχανισμό προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα. Όπως είπατε, και εσείς υπάρχουν, ε, υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση των ε, προτάσεων που έχουμε και να σας επιστήσω την προσοχή σε κάποιες από αυτές. Ε, νομίζω πως η επιβολή δασμών στα σύνορα δεν θα βοηθήσει το περιβάλλον, ούτε θα το προστατεύσει. Το μόνο που θα κάνει είναι να ενεργήσει προς όφελος των επιχειρήσεων, κάποιων επιχειρήσεων ίσως. Ε, θα μπορούσε ίσως να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός ανταμοιβή των ε, επιχειρήσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, είτε στην Ευρώπη είτε αλλού. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πιο καθαρή βιομηχανία σε σχέση με άλλες περιοχές και αυτό πρέπει να ανταμοιφθεί. Έπειτα με την, με την τροποποίηση ε, των, συντελεστών ΦΠΑ έτσι ώστε να μην γίνονται διακρίσεις στα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, είναι αυτές οι προτάσεις σύμφωνες με τους κανόνες του ΠΟΕ. Έπειτα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ETS και την χορήγηση πιστοποιητικών σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα, όπως ε, το ISO για παράδειγμα, τι γίνεται εκεί. Μετά, η ίχνη διαδικασιών όπως το blockchain. Ε, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Μπράβο σας, μπράβο σας. Τελευταίος ε, ο κύριος Εβαν Φόιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν οι πολίτες και αυτή η πράσινη συμφωνία είναι μία πολύ φιλόδοξη και σφαιρική απάντηση στις νόμιμα αιτήματά τους για δράση. Και είπατε προηγουμένως τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Ευρώπη. Η Πράσινη Συμφωνία λοιπόν είναι μία ελπίδα την οποία δεν θα πρέπει να την οποία δεν θα πρέπει να του απογοητεύσουμε, να μην δημιουργήσουμε απογοητεύσεις. Πρέπει όλοι μαζί να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την Πράσινη Συμφωνία. Η ερώτησή μου αφορά το μηχανισμό τον άνθρακα στις ε, παραμεθόριες περιοχές. Θέλω κάποιες λεπτομέρειες. Βάσει ποιων κριτηρίων κάποιοι ε, τομείς ε, θα υπαχθούν σε αυτό τον μηχανισμό, ποιοι θα αποκλειστούν. Θα πρέπει ο καθένας να ε, δηλώνει τα προϊόντα και τα ποσοστά για να ξέρουμε πού πηγαίνει. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα κονδύλια για αυτό το μηχανισμό και για το καλό των ε, ε, δικών μας των επιχειρήσεων. Θα ήθελα αυτά τα λεπτά να δίδονται μέσω του τμήματος έρευνας που θα την ανάπτυξή τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εάν ε, όταν διαφωνώ με την Λάγκε, διαφωνώ. Εδώ όμως συμφωνώ πρέπει να υπάρχει πλήρης παρερμηνία, διότι αυτό το οποίο είπα είναι ότι η ΚΑΠ οδήγησε στους γεωργούς το να ε, πιστεύουν ότι τους θεωρεί όλος ο κόσμος δεδομένους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό προσπάθησα να πω. Θα πρέπει λοιπόν να άρουμε αυτή την... Ε, ε, παρανόηση. Διότι θα πρέπει σε αυτή τη νέα κοινωνία που θέλουμε να κάνουμε, ουδέτερη από άνθρωπο, να τους... Ε, ε έχουμε στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να συμμετέχουν για να μπορέσουμε να έχουμε διαφορετική γεωργία και ασφαλή διαθροφή. Δεν ξέρω πώς δημιουργήσει η παρανόηση, αλλά κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Τώρα, ε, οι κρατικές ενισχύσεις. Ναι, ναι, θα το ξαναδούμε το όλο θέμα. Ναι, θα πρέπει να ε, δώσουμε κίνητρα στις ε, πράσινες επενδύσεις. Οι κανόνες για τις κρατικές επενδύσεις, για τις κρατικές επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο προευλέφθη τα πρέσια των κανονισμών έγινε πριν από την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα ε, περνάμε σε άλλο κύκλο θα πρέπει να δούμε αν κάποιοι από αυτούς τους κανόνες μπορούν να ισχύουν στην νέα αυτή εποχή που θα ζήσουμε. Ίσως όλοι να μην είναι κατάλληλοι. Ε, ε, όταν κάναμε τους κανόνες ε, δεν σκεφτήκαμε ότι κάποιοι θα πλουτίσουν υπερβολικά από την εφαρμογή τους κάποιοι όλοι. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα Δηλαδή θα πρέπει Ε, να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η πολιτική μας. Δηλαδή, δίνει κάποιος ελεύθερα τα δεδομένα που κατέχει κάποιοι τα χρησιμοποιεί, ε, στα, εμπορεύεται και πλουτίζει. Θα πρέπει λοιπόν να το ε, δούμε αυτό. Και έχω μία προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε περαιτέρω ε, φορολόγηση για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εάν τα κράτη που έχουν περισσότερα χρήματα και βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση ε, θα Εποφεληθούν περισσότερο από άλλα. Θα είμαστε λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην κάνουμε κάτι το οποίο θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα την Ευρώπη. Γι' αυτό λέγω ότι πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τύχουν μια της μελέτη αντικτύπου. Τώρα, για το μηχανισμό το άνθρακα στις ε, περιοχές. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε μορφή θα μπορούσε να είναι ε, αξιόλογη και αξιόπιστη για, την, για το αποτύπωμα των προϊόντων. Πώς το κάνετε αυτό και πώς οι διάφοροι παραγωγοί θα μπορέσουν αναπροϊόν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ειλικρινά θα πρέπει να φτάσουμε σε μια φάση στην οποία θα ελέγχουμε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθηθούν και οι δημόσιες αρχές και οι καταναλωτές θα είχαν, εάν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται για κάθε προϊόν και αν δούμε σε ποιο ποσοστό αυτό επηρεάζει την τιμολόγηση των προϊόντων και την ανταγωνιστικότητα. Εάν μπορέσουμε να κάνουμε ε, χάλιβα στην Ευρώπη με ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας αντί να χρησιμοποιούμε τα ορυκτά καύσιμα και είναι πιο φτηνά και είμαστε πιο ανταγωνιστικοί με τους άλλους και όλα γίνονται με τους σωστούς κανόνες τόσο το καλύτερο. Άρα θα πρέπει να γίνει η διόρθωση της τιμής ε, ώστε να είναι ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα μας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει, όπως σας είπα, με την διόρθωση. Πρώτα απ' όλα, ορίζοντας τα προϊόντα, βλέποντας ποια είναι η φορολόγηση των πρωτιών, με χρησιμοποιούμε τις μεθόδους ETS, αλλά πρέπει ούτως ή άλλως να είμαστε πραγματιστές. Θα συμβεί κάτι τέτοιο με κάποιο τρόπο, διότι εμείς... Ε, Πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να σταματήσει να είναι ευάλωτη η οικονομία μας. Τώρα, για το συμπληρωματικό κόστος για τους καταναλωτές. Θα έλεγα, ας προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε ενδεχομένως το συμπληρωματικό κόστος δράσης με το συμπληρωματικό κόστος αδράνειας. Μη ανάληψης δράσης. Και νομίζω ότι στη συγκέντρωση των δημάρχων που έγινε στην Βαρσοβία, στην Πράγα, στην ε, και στις, διπλο, στις ε, γειτονικές τους χώρες ήταν πραγματικά μια κραυγή για να κάνουμε κάτι να αλλάξει η ρήπα του περιβάλλοντος, ο αέρας, η κακής ποιότητας αέρας. Θα πρέπει, όπως ξέρουμε, να καταπολεμήσουμε τους πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη που είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εξαιτίας ε, του βεβαρημένου κλίματος στο οποίο ζουν. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν. Και πιστεύω ακράδαντα ότι το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί εάν βοηθήσουμε τα άτομα να κάνουν καλά μονομένα κτίρια, εάν ζουν σε υγιή κτίρια αν χρησιμοποιήσουμε το, την ξυλία για να κάνουμε και πιο οικολογικά σπίτια αν θέλετε. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε μετάβαση γίνεται με κόστος και συμπληρωματική δυσκολία, αλλά τα ωφέλη είναι επίσης τεράστια. Φανταστείτε πόλεις πράσινες, εγκαταλείποντας πλήρως τον άνθρακα πόσο πιο ελκυστικές θα γίνουν, πόσο πιο υγιείς και το κόστος δημόσιας υγείας θα πέσει πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Επίσης πιστεύω και εδώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε, να ξεχάσουμε κανέναν. Σε κάποιες περιοχές η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλους. Έχουμε κράτη-μέλη στις οποίες πίεση, τουλάχιστον το μισό ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιείται είναι ανανεώσιμη. Στην Πολωνία το 80% της ενέργειας προέρχεται από τον άνθρακα και θα πρέπει ε, κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Το έχουν καταλάβει οι Πολωνοί. Πρέπει να απαλλαγούν από αυτή την εξάρτηση από τον άνθρακα. Το καταλαβαίνουν. Και λέει η κυβέρνηση, αν πρέπει να το κάνουμε, θα το ε, πρέπει, ε, αν θέλετε να το κάνουμε με το ρυθμό που θέλετε, θέλουμε αλληλεγγύη, θέλουμε τη βοήθειά σας. Και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να είναι η μετάβαση δίκαια. Ναι, αλλά αυτό το ταμείο ε, μόνο με 100 εκατομμύρια τι μπορεί να κάνει. Ακούστε, προς το παρόν Α τα αφήσουμε έτσι και αργότερα θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά θα επανέλθω σε εσά όταν θα έχω πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Επίση, θα πρέπει να δώσουμε και νέα κατεύθυνση στα νέα μέτρα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μα. Δεν είναι το μοναδικό ταμείο αυτό, αλλά θα πρέπει αυτό το ταμείο και αυτή η πολιτική γενικότερα της αλλαγής να υποστηριχθεί και από όλα τα άλλα κοινοτικά ταμεία και κονδύλια που έχουμε. Έτσι θα δημιουργήσουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για να δώσουμε και κίνητρα στα κράτη-μέλη να αλλάξουν την πολιτική τους και να δώσουμε και κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δαπανούμε τα κονδύλια μας. Τώρα, όσον αφορά τα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου υπουργών. Α, έφυγε ο συναδελφός σας. Το αφήνω για άλλη φορά. Τώρα, είπα κάτι για το ταμείο και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Μιλούμε για διόρθωση αδικιών. Και το να διορθώσουμε τα πράγματα σημαίνει ότι κάνουμε μία διόρθωση, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα ε, κοινωνικά τα οποία θα πρέπει να δούμε και υπάρχουν και κάποιες ε, βιομηχανίες που θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο. Τώρα, σαν αφορά τη γεωργική παραγωγή, είπα αρκετά στην, πρώτη, στην απάντηση των πρώτων ερωτήσεων, πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Αυτό σημαίνει απαραίτητο ότι θα πρέπει να έχουμε λιγότερα ε, ζώα, λιγότερη κτηνοτροφία. Όχι απαραίτητο. Κάποιοι κάνουν ήδη μια τέτοια επιλογή, είναι δικό τους θέμα. Αλλά δεν κάνουμε αρκετές επενδύσεις στα ε, ζωοτροφές που δημιουργούν λιγότερες ε, εκπομπές. Λένε ότι είναι οι κτηνοτρόφοι τέτοιου είδους ζωοτροφές πιο δαπανηρές αλλά ο καθένας θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και να αναλάβει τις ευθύνες του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά με τον αγροτικό κόσμο και τον αγροτικό τομέα, όχι κατά των αγροτών. Αυτό το λέω και το υπογραμμίζω. Χρειαζόμαστε τους γεωργού περισσότερο από όσο ποτέ στα πλαίσια αυτή της πατάβαση. Αλλά θα πρέπει να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε διαφορετικά τα πράγματα. Να κάνουμε προτάσεις και να μην θεωρούμε ότι είναι στην ε, απέναντι πλευρά εχθροί μα. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε. Για τη διαχείριση των δασών η αναδάσωση δεν είναι η απάντηση για την αποψήλωση των δασών, δεν είναι η απόλυτη απάντηση, αλλά είναι, πρέπει να γίνεται σωστά παρόλα αυτά. Ο δικό μα ρόλο είναι να δώσουμε τα καλύτερα δυνατά επιστημονικά στοιχεία, ώστε να μην γίνουν σημαντικά λάθη στην αναδάσωση. Αλλά δεν μπορεί η αναδάσωση να αποτελεί μια δικαιολογία για να παραβλέπουμε την αποψήλωση των δασών ή η εξαφάνιση ε, του δάσου των τροπικών δασών δεν μπορεί να ε, καλυφθεί με την αναδάσωση. Και η επισήμανση, συμφωνώ, δεν είναι η απάντηση μόνη τη, είναι κομμάτι τη απάντηση. Είναι μία λύση. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε όλη την αλυσίδα παραγωγή και διανομή. Εδώ η εκτίμηση αντικτύπου μπορεί να έχει μεγάλη χρησιμότητα γιατί μπορεί να υπολογίσει το κόστο και το αποτέλεσμα τη επισήμανσης ε, με την εκτίμηση αντικτύπου. Είναι κομμάτι τη λύση, τόσο θεωρώ, όχι όλη η λύση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι χώρε ε, όπου γίνεται παραγωγή ε, προϊόντων που εξάγονται στην Ευρώπη θα αλλάξουν τη στάση τους και θα προχωρήσουν σε αναδάσωση και θα εκλείψει εκεί η αποψήλωση δάσεων, όχι αντιθέτως. Ε, συμφωνώ λοιπόν με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ναι, λοιπόν, η Κομισιόν αποφάσισε και το ανακοινώσαμε στην Πράσινη Συμφωνία ότι θα είμαστε πιο στήρι στην ε, εφαρμογή. Δεν έχει ακουστεί το μήνυμα παντού, αλλά θα πρέπει. Ναι, θα είμαστε πιο αυστηροί με την επιβολή, με την εφαρμογή. Ταυτόχρονα αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, διότι για παράδειγμα για τη δασοκομεία η μόνη δύναμη που έχουμε είναι η δύναμη τη πυθού. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε σχέδια τα οποία θα μα βρίσκουν συμφωνού όλου. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι. Τέλος, ε, στην τελική ερώτηση θα δούμε και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τις ξαναδούμε. Πράγματι η βιομάζα, η πλάνη, ότι οτιδήποτε έχει τη λέξη βίο μπροστά του είναι καλό, πρέπει να μην ε, την πιστεύουμε. Η βιομάζα δεν είναι από μόνο της καλή. Πρέπει να βλέπει κανείς τι ποιότητα έχει η βιομάζα αν αρχίσουμε να φτιάχνουμε πέλετσε και να τα καίμε σε τεράστιε ποσότητες αντί για κάρβουνο, δεν είμαι τόσο βέβαιο ότι συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πολύ. Και επίση όσον αφορά την αναδάσωση, αν πάμε να κάνουμε αναδάσωση για να καλύψουμε, ε, για να καλύψουμε το ότι κόψαμε δέντρα 100 ετών, δεν είναι βέβαιο ότι κάνουμε σωστά, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά. Απάντησα ήδη για την ε, ένταση άνθρακα και για το μηχανισμό προσαρμογής των άνθρωπων στα σύνορα. Αυτά, συγγνώμη. Αυτά. Thank you for this, uh, Ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ξανασυναντηθούμε του χρόνου, 13 Ιανουαρίου. Καλά Χριστούγεννα, καλές διακοπές.